So, good morning everybody. It's a pleasure welcoming you. Καταλαβαίνω ότι βέβαια το Βέλγιο δεν είναι τόσο ευχαριστημένο σήμερα. Δεν βλέπω Γάλλους αδέλφους, φαίνεται ότι ορτάζουν ακόμη. Και οι Βρετανοί προετοιμάζονται. Και οι Κροάτες το ίδιο. Έγκριση μερίσας διάταξης. Παρατηρήσεις? Όχι. Ανακοινώσει του Προέδρου. Έχω ορισμένε. Πρώτα απ' όλα συστάσεις ε, των συντονιστών. Μετά τη συνεδρίαση των, ε, της 20ης MFF, η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιτροπών, ο κανονισμός ε, για τις κοινέ προβλέψεις θα ε, ασκήσουμε το άρθρο 54 αποκλειστική αρμοδιότητα για το άρθρο 15. Επίσης, είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε το κανόνα 53 συν ανταγωνιστικότητα, ε, ενιαία αγορά και ευρωπαϊκές στατιστικές. Είπαμε ότι θα αποσταλεί, ε, αποσταλεί επιτροπή α, επιστολή, εκονήτρε γιατί αυτές είναι οι επιτροπές οι οποίες ενδιαφέρονται περισσότερο. Και η διάσκεψη των Προέδρων συμφώνησε ότι το οίκον θα πρέπει, η οίκον θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την διαδικασία αυτή διορισμοί. Ο διορισμός για τον μηχανισμό κατά της απάτης για το για το ε, ΦΠΑ πήγε στο ΕΛΚ για τα ενοπνευματώδη ΚΟΕ παρακολούθηση των ε, ε, ειδών πολυτελείας δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει γενική γενικός κανονισμός για τα προϊόντα πολυτελείας ΓΚΟΕ, συνεργασία για τα ηλεκτρονικά μητρώα EPP, εισαγωγή των τεχνικών μέτρων για το τελικό σύστημα ΦΠΑ για τη φορολόγηση του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών ΕΛΚΕ, δημιουργία του συστήματος για την αναθεώρηση ε, της ε, στήριξης, ε, ALDE, ε, δημιουργία ενός ευρωπαϊκού, ε, μιας ευρωπαϊκής λειτουργίας ε, συστήματος σταθεροποίηση των επενδύσεων, S&D, συνεργασία στον τομέα του φυσκάλης πράσινη, η, τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ορισμένες κατηγορίες ε, οριζοντίων ε, κρατικών επιδοτήσεων, ECR, πρόταση για κανονισμό του Συμβουλίου που να τροποποιεί τον κανονισμό 1553 89 για την οριστική ρύθμιση για τη συλλογή ιδίων πόρων από το ΦΠΑ. Δεν θα γνωμοδοτήσουμε γι' αυτό. Πρόταση για μια απόφαση του Συμβουλίου για το σύστημα ιδίων πόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση Σοσιαλιστέ. Μείωση τη επίπτωση ορισμένων πλαστικών στο περιβάλλον, ENF. Κοινέ ε, διατάξει του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου, του Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για, τις, για την αλληλεία και τις θάλασσες και οι οικονομικοί κανόνες για το Ταμείο για το άσυλο, την εσωτερική ασφάλεια, τη διαχείριση των συνόρων και τις θεωρήσεις πηγαίνει στο ΕΛΚΑ. Ωραία. Εφόσον το, ε, η διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει για τις αρμοδιότητες. Η πρόταση για ένα κανονισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάρριξη των κανονισμών, διαφόρων κανονισμών. Δεν θα τις διαβάσω. Στο ECR και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για, την για την, το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής και η ετήσια έκθεση ανάπτυξης 2019 θα πάει στο ΕΛΚ. Για τον Brexit δεν έχω βλέπω τίποτα. Οι αντιπροσωπείς μας για το δεύτερο εξάμεινο Κίνα, οι συντονιστές ενημερώθηκαν ότι η Επιτροπή Οικονομικών του Κοινοβουλίου της Κίνας επιβεβαίωσαν θα πάμε το Σεπτέμβριο. Οι συμμετέχοντες θα είναι ως εξή. Για την Κίνα, τρει ΕΛΚ, τρει σοσιαλιστές μαζί με τον πρόεδρο, ένα ΣΥΣΙ, ένα ΣΑΛΤΕ. Η ετήσια συνάντηση του Διεθνούς Ομοσπονδιακού Τμήματος στον Πάλι, τρει ΕΛΚ, τρει σοσιαλιστές με τον πρόεδρο, ένα ΣΥΣΙ, ένα ΣΑΛΤΕ και Ιταλία, 4 ΕΛΚ, 4 ε, σοσιαλιστές μαζί τον πρόεδρο, Ένα CCR και ένας ΑΛΤΕ. Οικονομική διακυβέρνηση. Οικονομικό διάλογο με τον Ισπανό Υπουργό Οικονομικών συμφωνήθηκε να τον προσκαλέσουμε σε ένα οικονομικό διάλογο το δεύτερο εξάμεινο το 2018. Και συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια για τι αναχώρα συστάσει, οι συντονιστέ επιβεβαίωσαν ότι θα λάβει η χώρα στι 9 Οκτωβρίου. Αναφορέ. Δεν έχουμε σχόλια για την πληροφόρηση που δόθηκε για την προφορική ερώτηση για το ΦΑΤΚΑ και το σχέδιο ψηφίσματος που έχει εκπονήσει η Επιτροπή Αναφορών. Και επίσης θα έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας για την EIB. Θα στείλουμε μια επιστολή στους προέδρους των επιτροπών ζητώντας να μας δώσουν δυνατότητα να κάνουμε αυτή την έκθεση. Αυτή είναι η συνήθιση διαδικασία και μια νομερημένη εκδοχή του προγράμματος επιστολή, της επίσκεψης στη Washington θα σταλεί στους συντονιστές μετά από τη συνεδρίαση. Ο Υπουργό Οικονομικών τη Βουλγαρία θα έρθει αύριο σε εμά για μία σύντομη παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων για το τέλος της Προεδρίας και μετά την ε, δημόσια συνεδρία 19 Ιουνίου είπαμε ότι θα υποβάλουμε μια πρόταση για την λάθος πώληση χρηματοπιστωτικών προϊόντων για την μη σωστή εφαρμογή του νόμου. Δεν υπήρξε αντίρρηση. για την ε, δήλωση του Προέδρου να μην γίνει συνάντηση με τους ε, συντάκτες έκθεσης. Ε, τώρα, γνωμοδότηση για τον νόμο για τις διεκδικήσεις. Δεν θα κάνουμε γνωμοδότηση Αυτό έχει ήδη Τώρα η επιτήρηση, μία επιστολή για το Φεργιώτα 2 θα αποσταλεί στην Επιτροπή και ο πρώην πρόεδρος ε, της Ελστατ, ο πρόεδρος είπε ότι θα στείλει μια επιστολή στους συντονιστέ για σχόλια και θα θίξει το θέμα κατά τη συνεδρίαση της ε, ομάδας ε, εργασίας για την οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα που έχει ήδη λάβει χώρα. Αυτά, αυτές οι ανακοινώσεις μου. Οι διερμηνείς θα αναλάβουν δράση σήμερα. Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρξει δερμηνία μόνο για τις, ε, είναι εγγυημένη μόνο για τις πέντε κύριες γλώσσες. Θα δούμε τι θα προκύψει. Να περάσουμε στο σημείο 3, παρακολούθηση των ε, έλεγχων των ε, κατεξοδότηση πράξεων και εφαρμοστικά μέτρα. Είναι 14η φορά που το κάνουμε αυτό δεν έχουμε τίποτα για να το γιορτάσουμε. Η εικόνα αποδίδει μεγάλη σημασία, ή στη 40 μάλλον, έχουμε μεγάλη, αποδίδει μεγάλη σημασία στη σημασία της αποτελεσματικής άσκησης αυτών των καθηκόντων. Θα ασχοληθούμε με τα μέτρα επίπεδου 2, ε, υπό τον κανονισμό BMR από την 1η Ιανουαρίου 2018. Οι περισσότεροι κανόνες για τις ε, τιμές αναφοράς δίνουν ε, στοιχεία με βάση ορισμένες τιμές αναφοράς, αλλά πρέπει να ε, εφαρμόσουμε ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές που θα συζητήσουμε σήμερα. Καλώς ορίζω τον κύριο Τίλμαν Λούντερ, που είναι επικεφαλής στην DG FISMA, επικεφαλής της μονάδας για τις ε, αγορές ε, μετοχών και αξιογράφων και τον κύριο Ιάκουμ Μιχάλη που επίσης είναι εκπρόσωπος του ΕΣΜΑ. Σας παρακαλώ να μας κάνετε μια σύντομη εισαγωγή, δεν θα πρέπει να κρατήσει πάνω από 5 λεπτά. Να ακούσουμε λοιπόν πρώτα την Κομισιόν και μετά θα μιλήσουν οι συνάδελφοι. Επιτροπή λοιπόν πρώτα, έσμα μετά και μετά ε, ο εισηγητής μας και οι Σκιώδης. Ο κύριος Λούντερ. έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Σήμερα Θέλουμε να σας παρουσιάσουμε 10 ε, ρυθμιστικές προδιαγραφές με βάση τον κανονισμό για τις τιμές αναφοράς που αφορούν την, ε, τον έλεγχο λειτουργίας, ε, τα στοιχεία που βάζουμε, τη μεθοδολογία, τη διαφάνεια. Το πιο σημαντικό νομίζω είναι ο κώδικας διοντολογίας για τους συμβάλλοντες και έχουμε και άλλα κριτήρια για τις σημαντικές τιμές αναφοράς. Έχουμε και τη δήλωση τιμών αναφοράς, η ρυθμίσει για τη συνεργασία και το σύστημα για την αναγνώριση των τρίτων χωρών. Όπως ξέρετε, αυτά είναι ιδιαίτερα τεχνικής φύσης, τα RTS. Είναι επιπλέον ε, έντυπα μετά τις ε, υποχρεώσεις που θέτει η πρωτογενής νομοθεσία. Η ΕΣΜΑ μας έστειλε όλες αυτές τις προδιαγραφές και θα τις εγκρίνουμε χωρίς καμία ουσιώδη αλλαγή. Οι αλλαγές που βλέπετε είναι απλώς ε, στις διατυπώσεις. Και κατά τη γνώμη μας δεν αλλάζουν την ουσία των τιμών αναφοράς της ε, ΕΣΜΑ. Αν δείτε ότι έχει αλλάξει κάποια διατύπωση, δεν αφορά την ουσία Βεβαίως όπου υπάρχουν ε, κάποια υπερβολικά προβλήματα, κάποιες φόρτος εργασίας, αυτό έχει να κάνει με το ότι θέλουμε να αλλάξουμε κάποιες διατυπώσεις, αλλά να βεβαιωθούμε ότι δεν θα αλλάξει ουσία. Αυτό μας πήρε κάποιο χρόνο. Αλλά η μεγαλύτερη καθυστέρηση που αντιμετωπίζουμε είναι ότι η μετάφραση αργεί έχουν φόρτο εργασία οι υπηρεσίε μετάφραση. Ναι, καθυστερούμε λοιπόν, είναι ευθύνη μα, το παραδεχόμαστε. Ε, κάνουμε έκκληση ε, για την επίοικια από πλευρά σα, γιατί οι μεταφραστικέ υπηρεσίε ε, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν, υπάρχει σημαντικό φόρτο εργασία. Είναι σημαντικέ προδιαγραφέ αλλά αποφασίσαμε να μην τους δώσουμε την ε, ύψιστη προτεραιότητα στο πρόγραμμα εργασιών της μεταφραστικής υπηρεσίας, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι στο επίπεδο 1 η πρωτογενής νομοθεσία είναι σαφής. Δεν θα κάνω άλλα σχόλια. Θα το αφήσω αυτό στο συνάδελφο της ΕΣΜΑ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, ε, κύριε Λούντε. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Μιχάλικ από την ΕΣΜΑ. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, σας ευχαριστώ που δίνετε στην ΕΣΜΑ την ε, δυνατότητα να συμμετάσχει στη συναντρίασή σας για τα μέτρα επίπεδου 2 του κανονισμού για τις δείκτες αναφοράς, PMR. Αυτό έχει σαν απότερο στόχο να φτάσουμε στους στόχους των συνομοθετών. Θα σας μιλήσω για αυτές τις δραστηριότητες. Η ΕΣΜΑ έχει υποβάλει 11 πρότυπα στις 30 Μαρτίου 2017 και επιπρόσθετα πρότυπα τον Ιούνιο του 2017. Σας δώσαμε το ε, περιεχόμενο ήδη στις 8 Ιουνίου του 2017. Επίσης υπάρχει μία εποπτεία και ένα εποπτικό πλαίσιο που δόθηκε στη Γραμματεία. Με βάση του στόχους του επίπεδου 1, τα επίπεδα σχετίζονται με την ε, ακαιρεότητα και την ευρωστία των μέτρων μέσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας έχουμε εισαγάγει την αναλογικότητα, ιδιαίτερα για τους διαχειριστές σημαντικών και μη δικτών αναφοράς, έτσι ώστε οι συνομοθέτες να έχουν ένα πιο λεπτομερές πλαίσιο που αφορά τους διαχειριστές η καθυστερημένη εφαρμογή του RTS θέτει σε κίνδυνο την εφαρμογή του κανονισμού BMR. Γι' αυτό η ΕΣΜΑ θα ήθελε η Επιτροπή να ε, εγκρίνει το RTS. Στη συνέχεια η ΕΣΜΑ ασχολήθηκε με τους δείκτες αναφοράς για να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός. Στα, επίπεδα, στα μέτρα του επίπεδου 3 η ΕΣΜΑ έχει ε, προωθήσει μέτρα, ιδιαίτερα για τους δείκτες αναφοράς ίσονος σημασίας στις 29 Σεπτεμβρίου 17. Θεωρούμε ότι αυτοί οι δείκτες θα πρέπει να αφορούν τον έλεγχο τα στοιχεία εισαγωγής, τη διαφάνεια μεθοδολογίας και την διαχείριση αυτών των στοιχείων. Το περιεχόμενο αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών σχετίζεται με αυτά τα τέσσερα σημεία. Γι' αυτό η ΕΣΜΑ αναμένει την ε, έκδοση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών στην επίσημη εφημερίδα των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, από τον Ιούλιο του 2017 προσπαθούμε να προωθήσουμε αυτή τη διαδικασία μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων έτσι ώστε να δουν όλοι πώς ισχύουν αυτές οι τιμές αναφοράς. Στόχος είναι οι επενδυτές και άλλες, άλλοι φορείς αγοράς να έχουν επιπρόσθετα μέτρα. Ε, Προσθέτω, την 1η Ιανουαρίου 2018 έχουμε το πρώτο ε, μητρό έσμα για τους ε, ε, διαχειριστές τρίτων χωρών και τη μόνο αναφοράς. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει ένα δίκτυο αναφοράς εάν περιλαμβάνεται στο μητρό. Το μητρό αυτό που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας έχει ήδη 14 διαχειριστές δυνάμει του κανονισμού BMR και θεωρούμε ότι αυτός ο αριθμός θα διπλασιαστεί πριν από το τέλος του έτους. Επίσης, τρεις δείκτες αναφοράς έχουν ήδη εγκριθεί, ε, Euribor, Αιώνια και Libor. Δύο συνάδελφοι των αρμοδίων αρχών ασχολείται με, ασχολούνται με την εποπτεία του Euribor και της αιώνια, ενώ ο δεύτερος ασχολείται ε, με το LIBOR με βάση τις, ε, ε, τα δεδομένα της Βρετανικής Αρχής Κινητών Αγορών. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε σύγκληση των πρακτικών εποπτείας και γι' αυτό το λόγο στις 2 Ιουνίου 2017 εγκρίναμε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο έτσι ώστε να δούμε ποιοι θα ήταν οι ενδυνάμοι υποψήφοι για τα υποχρεωτικά μέτρα και τιμές αναφοράς το Φεβρουάριο του 2018 η ΕΣΜΑ μαζί με την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροφή, Επιτροπή καθώς και τις Βελικές Αρχές ε, όρισε μία ομάδα εργασίας έτσι ώστε να εξευρεθούν εναλλακτικοί ε, δείκτες χωρίς κίνδυνο. Επίσης, έχουμε εκινήσει μια διαδικασία διαβουλεύσεων στις 21 Ιουνίου 18 για εναλλακτικούς δείκτες και ενδυνάμει υποψηφίους. Επίσης, αυτό που μας ενδιαφέρουν είναι δύο δείκτες δανεισμού και οι συγκεκριμένοι δείκτες και επιτόκια βραχυχρόνιου δανεισμού. Σας ευχαριστώ πολύ και παραμένω στη διάθεσή σας για να απαντήσω οποιασδήποτε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα το ε, έχει η Καρολίνα Ντεγκάρ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την ε, Επιτροπή ε, που μας έδωσε πληροφορίες για, τις, για τους δείκτες αναφοράς. Θεωρούμε ότι οι αρμόδιες αρχές τώρα ασχολούνται με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας και των σχετικών δικτών αυτό το νέο καθεστώς θα επιτρέψει την άμεση εφαρμογή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τρίτες χώρες ως προς τους δείκτες αυτούς αναφοράς. Μετά από έξι μήνες θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τα μέτρα εφαρμογής έτσι ώστε όλοι να συμμετάσχουν. Το πρώτο σημείο αφορά τον ίδιο τον κανονισμό, BMR. Μιλάμε για τα μέτρα αυτά που έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή, ε, στην Επιτροπή από την ΕΣΜΑ τον Ιούνιο του 2017, δηλαδή πρόκειται για ένα χρόνο πριν και άρα βρισκόμαστε σε μία περίοδο μετά το αρχικό τρίμηνο που προβλεπόταν. Έχουμε μία επεξήγηση από την Επιτροπή, αλλά θα ήθελα να πω ότι δεν δέχομαι αυτή την καθυστέρηση. Ε, ιδιαίτερα σε σχέση με την παροχή των δικτών αναφοράς. Δύο εβδομάδες πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έδωσε ένα ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο έτσι ώστε να το αναλύσουμε. Θεωρώ ότι τα μέτρα που πρότεινε η ΕΣΜΑ είναι περιορισμένα. Η προσέγγιση όμως της Κομισιόν είναι ακόμα πιο συσταλτική Δηλαδή στο άρθρο 1 αναφέρει αντί περιλαμβάνονται το considered to include. Ελπίζω η Επιτροπή να ε, μας πει για ποιο λόγο θα γίνει η εκτέλεση, εκτέλεση των μέτρων δύο μήνες μετά τη θέση σε εφαρμογή. Σε σχέση με το, τα, τους δείκτες αναφοράς στα πλαίσια του ρυθμιστικού ε, εντύπου θα πρέπει να ορίζονται από το άρθρο 3 συμπεριλαμβάνοντας τις λέξεις entirely and directly. Αυτή η συσταλτική ερμηνεία του κειμένου επίπεδου 1 θα μπορούσε να βρεθεί εκτός πλαισίου ρύθμισης των δικτών αναφοράς και θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές επειδή υπάρχουν περιορισμένοι δείκτες αναφοράς. Αυτό δεν αντικατοπτρίζει την αναλογικότητα των προαπαιτήσεων για διαφόρους δείκτες αναφοράς μετά από συμφωνία στους τριμερείς θα θέλαμε να αρχίσουν οι συζητήσεις για το πώς μπορούν να εξευρεθούν λύσεις για να μην υπάρξει νομική ασάφεια και ανασφάλεια. Θεωρούμε ότι οι, οι ρυθμιστικοί αυτοί δείκτες αναφοράς θα πρέπει να ορίζουν την αγορά μέσα στα πλαίσια και του MIFID 2. Έτσι, η ποιότητα των στοιχείων είναι αδιαμφισβήτητη και μπορούμε να δράσουμε εάν υπάρχουν απάτες. Θεωρούμε ότι οι αλλαγές του επίπεδου 1 είναι και οι πλέον επιθυμητές μέσα στα πλαίσια αυτής της ολοκληρωμένης προσέγγισης και ακαιρεότητας θεωρώ ότι οι συνομοθέτες, οι αποκοινού νομοθέτες θα μπορέσουν να συνεργαστούν μέσα στα πλαίσια των ρυθμισμένων δικτών αναφοράς και μπορούμε να έχουμε ένα οριστικό πλαίσιο τους επερχόμενους μήνες. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μία αναθεώρηση μέσα στα πλαίσια του συνολικού πακέτου που διέπει τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Θα πρέπει να είναι δυνατόν να δώσουμε τελική μορφή σε αυτούς τους δείκτες πριν από την 1η Πρώτου 2020. Εάν ε, δεν δοθεί οριστική μορφή σε αυτούς τους δείκτες αναφοράς, θα ήθελα η ΕΣΜΑ να χρησιμοποιήσει ό,τι ε, μέσο έχει στη διάθεση της για να βρούμε μία λύση σε επίπεδο 1 έτσι ώστε να, λα... να ληφθούν υπόψη οι προθέσεις των ε, αποκοινού νομοθετών για να υπάρχει σταθερότητα στις αγορές. Ελπίζω οι συνάδελφοι και η Επιτροπή να υποστηρίξουν αυτή την προσέγγιση. Επίσης, με απασχολεί το θέμα της μετάβασης του Euribor και της αιώνια Νομίζω ότι λήγουν οι προθεσμίες στην πρώτη η πρώτη πρώτου 20 και μέχρι τότε μπορεί να έχουμε εναλλακτικέ για την αιώνια. Επίσης υπάρχει μεγάλη ε, αμφιβολία και ανησυχία σε σχέση με την μετάβαση και αναθεώρηση του ε, επίπεδου που αφορά τη Euribor, τι θα γίνει σε περίπτωση ε, αναστάτωσης της αγοράς. Θεωρώ ότι θα έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία σε σχέση με τα θέματα τα οποία εκκρεμούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Καρολέν και από το ΕΛΚ το λόγο έχει ο κύριος Ταρούς Ροζάτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφο, ο Σκιώδη από το ΕΛΚΑ δεν μπορεί να παραβρεθεί σήμερα και ζητά συγγνώμη για την απουσία του αυτό και με ζητά να ενημερώσω την Επιτροπή αυτή ότι χωρί περαιτέρω παρατηρήσεις υποστηρίζει ε, την εισηγήτρια και συμφωνεί με τα σχόλια που έκανα. Θα ήθελα να ευχαριστήσει ιδιαίτερω επίση την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε σε αυτό το πολυτεχνικό φάκελο, τον οποίο και κληρονόμησε από την προηγούμενη η συγκητρία την κόρα Φαν και τη έφυγε κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντάριο. Και να περάσουμε στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο Χων Φερνάντε. Ευχαριστώ. Έχει περάσει αρκετό χρόνο. Το είπε ο εκπρόσωπο τη ε, Κομισιόν. Μα πήρε πολύ χρόνο η εκπόνηση των, διαφόρων ε, νομισματικών μέτρων που έπρεπε να πάρει η Κομισιόν και η ΕΣΜΑ. Τρία χρόνια περιμένουμε για να εγκριθεί αυτό το κείμενο από τους συνομοθέτες. Στις αρχές του 2014, όταν ε, κατέβηκα σε ευρωεκλογέ, ήταν περίπλοκη η κατάσταση, όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά παντού στην Ευρώπη. Υπήρχε μια οικονομική και τραπεζική κρίση πολύ σκληρή, αλλά ε, υπήρχαν και κακές πρακτικές πολλών πιστοτικών ιδρυμάτων που είχαν ε, επηρεάσει και είχαν εξαπατήσει και τελικά είχαν ε, αποσπάσει πόρους από τους καταθέτες και επενδυτές με πρακτικές που ήταν αντίθετες με την νομοθεσία και γι' αυτό χρειαζόταν ένας κανονισμός για να υπάρχει μια διαφανής διακυβέρνηση, μια σωστή διακυβέρνηση με σωστούς οικονομικούς δείκτες, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε καμία ρύθμιση για όλα αυτά τα πιστοτικά ιδρύματα. Κατέβηκα σε ευρωεκλογέ ε, λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να γίνονται ε, ενέργειες για τον επηρεασμό του Euribor, του Libor, όλα αυτά τα οποία είχαν ε, οδυνηρές επιπτώσεις για τους πολίτες Ευρώπης. Έπρεπε να τελειώσουν όλα αυτά. Υπάρχει μία ρύθμιση για να αποφεύγονται τέτοια θέματα. Αυτό το θέμα συζητήθηκε και από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο και σε λιγότερο από ένα χρόνο κατέληξαν τα δύο όργανα σε συμφωνία, καλή συμφωνία που θα ελαχιστοποιούσε ή θα καταργούσε τη δυνατότητα των πιστοτικών ιδρυμάτων να επηρεάζουν τόσο σημαντικούς δείκτες όπως το Euribor και το Libor. Αλλά βλέπουμε ότι μετά από τόσα χρόνια δεν εφαρμόζονται όλα αυτά. Θέλουμε υπερβολικά πολύ χρόνο για να εφαρμόσουμε, για να εκπονηθούν μάλλον οι διάφορες ε, κατεξοδότηση πράξη και οι τυπικές διαδικασίες. Και υπάρχει και αντίσταση από τον τομέα. Πρέπει να το πούμε. Δεν θέλουν να εφαρμόζουν ε, αυτά που προβλέπουν αυτά τα κείμενα. Το βλέπουμε και τώρα με το Λίμπορ. Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και όλοι οι άλλοι οργανισμοί επίβλεψης δεν πρέπει να συνεχίσουν να ανέχονται αυτή την κατάσταση. Οπότε, τονίζω, εφόσον έχουμε τώρα διαδικασία ελέγχου, ότι πρέπει να βιαστούμε για να υπάρξει η εφαρμογή των αποφάσεων. Ούτω ώστε αυτοί οι κανόνες να εφαρμοστούν. Υπάρχει συγκεκριμένα ένα άρθρο για τις τιμές αναφοράς με τα ε, σωστά στοιχεία. Υπάρχουν κάποιες ε, αφιβολίες για το τι περιέχει τελικά το κείμενο που εγκρίναμε. Θεωρώ ότι επειδή αυτές οι τιμές αναφοράς τελικά εξαιρούνται από κάποια κριτήρια, αυτό οφειλόταν στο ότι αυτές οι τιμές αναφοράς που βασίζονται σε στοιχεία που ήδη ελέγχονται θα, μπορούσε να, θα μπορούσαν ακριβώς αυτές οι τιμές αναφοράς να, έχουν, να βασίζονται σε λιγότερες προδιαγραφές. Αλλά αυτές οι, οι τιμές αναφοράς. Μιλάμε για τιμές αναφοράς που βασίζονται σε τιμές αναφοράς. Εδώ μπορεί να υπάρξει επηρεασμός. Ενώ στο κείμενο λέγεται ότι τα, στοιχεία, τα στοιχεία πρέπει να παρέχονται από ε, έναν οργανισμό που να ελέγχεται. Και αυτή είναι η ουσία της ρύθμισης. Οι τιμές αναφοράς μπορούν να ελέγχονται λιγότερο. Αλλά αυτό που συζητάμε είναι τιμές αναφοράς που βασίζονται σε άλλες τιμές αναφοράς. Εδώ ήδη υπάρχει ενδεχόμενο επηρεασμού. Άρα εδώ πρέπει να υπάγονται σε όλους τους κανόνες που προβλέπει ο κανονισμός. Δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορεί να υποστηριχθεί ότι αυτές οι νομικές αμφιβολίες μπορούν να είναι παραθυράκι. για να επιτραπεί μαζική χρήση του κανονισμού για ε, τα benchmark που βασίζονται σε ελεγχόμενα στοιχεία. Του χρόνου έχουμε ευρωεκλογέ. Ελπίζω και επιθυμώ να μπορώ να πω στους Ισπανούς ε, πολίτες ότι δεν επηρεάζονται το Euribor, το Libor, ε, οι τιμές των πρώτων υλών και ελπίζω αυτές οι αμφιβολίες για την εφαρμογή του κειμένου να αντιμετωπιστούν σύντομα. Γιατί νομίζω ότι είναι πολύ απλό να επιληθούν. Εάν πραγματικά σεβαστούμε το πνεύμα του κειμένου. Σε ευχαριστώ και δεν βλέπω κανέναν άλλο από το ECR, ούτε από τους πράσινους να ζητάει το λόγο, ούτε και από την ΚΟΕ. Από το EFT, από το ENF, κανείς δεν έχει ζητήσει το λόγο. Επίσης, στη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΙ δεν έχουμε κανέναν. Και θα περάσουμε λοιπόν πάλι στα θεσμικά όργανα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε να πάρετε το λόγο και ύστερα από την ΕΣΜΑ. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ακούσαμε κάποιε ερωτήσει, τι οποίε και θα επιχειρήσω να απαντήσω. Νομίζω ότι πιο σημαντική ήταν ε, όντω το θέμα για τα, τους, τις τιμές αναφοράς ε, τις ρυθμιστικές. Το έχουμε υπόψη μας το θέμα αυτό και έχουμε κάνει και κάποια έρευνα, το έχουμε συζητήσει άλλωστε και στον 7ο τριμερή διάλογο για τη διαδικασία καθορισμού των τιμών αναφοράς στα τέλη του 2015 και πράγματι. Τότε ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήμανε ότι θέλει να διευρύνει το πεδίο της, ε, του ορισμού προκειμένου να περιλαμβάνει και διαμεσολαβητές οι οποίοι μπορούν να, μπορούν να έχουν πρόσβαση στα, στα δεδομένα αυτά. Το Συμβούλιο ήταν αντίθετο τότε γιατί θεώρησε ότι οι διαμεσολαβητές δεν ήταν ρυθμιζόμενε οντότητες και ως εκ τούτου ενδεχομένω στη φάση αυτή να υπήρχε χειραγώγηση σε ό,τι αφορά δηλαδή τους διαμεσολαβητές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να βρει μια μέση λύση και δήλωσε ότι σε κάθε περίπτωση αυτή οι διαμεσολαβητές στις πιο πολλές περιπτώσεις θα ήταν APAs, και φυσικά, αν τα στοιχεία αυτά προκύψουν άμεσα από έναν διαπιστευμένο βοηθό EPA, θα ίσχυαν τι ίδιε αρχέ. Άρα, αν δεν ρυθμίζεται αυτό από τη ρυθμιζόμενη αγορά, το οποίο ήταν το πιο αυστηρό κριτήριο, το οποίο και υποστήριζε τότε το Συμβούλιο, είπαμε ότι αν υπάρχει διαμεσολαβητή, ο διαμεσολαβητή ο ίδιο θα θεωρείται αμα, μία πηγή νόμιμη για την παροχή δεδομένων. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτός ο συμβιβασμός ακόμα αξίζει τον κόπο να εξεταστεί. Θυμόμαστε και τι είχε γίνει στον τρομερή διάλογο, υπήρχε κάποιο σκεπτικισμό σε ό,τι αφορά την χειραγωγήση στοιχείων και δεδομένων από τους ε, διαμεσολαβητές, ιδιαίτερα αν ήταν από πολλές πηγές τα δεδομένα αυτά. Από την άλλη, αν υπάρξει αλλαγή σε επίπεδο 1, σίγουρα θα το θεωρήσουμε και αυτό μια χρήσιμη εξέλιξη. Απλά σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει μια κάποια, ένα κάποιο ιστορικό πριν από, πίσω από το θέμα των διαμεσολαβητών και ότι τα στοιχεία αυτά των διαμεσολαβητών προέρχονται ήδη από ρυθμιζόμενες αρχές, χωρίς να παρεμβαίνουν στην διαδικασία μη διαπιστευμένη φορείς. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους APAs, τους διαπιστευμένους αυτούς ε, διαμεσολαβητές. Θα δούμε στην πορεία όμως πώς θα διαμορφώσουμε το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα την διαδικασία εποπτείας, τέθηκε η απέτηση να υπάρχουν εκπρόσωποι και από άλλες ε, οντότητες ε, που παρέχουν καθαρές ε, αξίες ως παρόχη. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό ως διαδικασία και άλλαξε όντω όσο, όπως επισήμανε και η συγκεκριά. Πιστεύω ότι θα πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθούν, γιατί πιστεύουμε ότι αποτελούν βασικοί, βασικούς φορείς και βασικούς εισφορείς Και άρα η ακυριότητα των δεδομένων τους θα πρέπει να εξασφαλίζεται. Θα πρέπει να συμμετέχουν λοιπόν και στο Συμβούλιο α, Διακυβέρνησης, γιατί παρέχουν α, ε, ακριβώς ε, τέτοιο ενεργητικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές αναφοράς αιώνια, όπως είπε η ΕΣΜΑ, υπάρχει μια κοινή ομάδα μεταξύ διάφορων θεσμικών οργάνων που συμπεριλαμβάνει και τον, τη Βελγική Ρυθμιστική Αρχή που είναι υπεύθυνη για την αιώνια, την ΕΣΜΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ομάδα εργασίας αυτής ακριβώς ε, εξετάζει εναλλακτικέ λύσεις και μέσα ε, ανευκινδύνου. Μία λύση λοιπόν ε, για να υπάρχει αυτή η ασφάλεια, αυτή η βεβαιότητα ή θα ήταν να λαμβάνουν δύο τιμές αναφοράς μια έγκριση. Έχουμε ακόμα χρόνο. Όπως επεσήμανε και η ΕΣΜΑ αλλά και η συγγήτρια, έχουμε ακόμα μια παραδοσιακή περίοδο ε, μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, άρα έχουμε χρόνο να επιλύσουμε το θέμα αυτό και να αποφύγουμε περαιτέρω διάβρωση των εισφορών μέσω Έγκριση των τιμών αναφορά. Αν αυτό τώρα δεν καταστεί δυνατό, θα έχουμε το θέμα ότι η μεταβατική περίοδο στην οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα χωρί έγκριση θα λήξει τον Ιανουάριο του 2020. Είμαστε λοιπόν τμήμα τη ομάδα εργασία αυτή και το παρακολουθούμε το θέμα αυτό. Σα υπενθυμίζω ωστόσο ότι έχουμε ακόμα και το υπόλοιπο 2018 καθώς και όλο το 2019 για να επιλύσουμε το θέμα αυτό. Ελπίζω δε και οι ρυθμιστικές αρχές που έχουν επιφορτωθεί με την έγκριση των τιμών αναφορά θα κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Από την άλλη, ασφαλώς, αν θα πρέπει να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα, φυσικά και θα δώσουμε καθοδήγηση και συμβουλές για το πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό χωρίς να υπάρχουν ζητήματα εφαρμογής. Σε περίπτωση που προκύψει, εν πάση περιπτώσει, ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί κάποιες, ε, κάποια από τις δύο αυτές τιμές αναφοράς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα να δώσω το λόγο στην Έσμα να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα, πάω πολύ, θα πω πολύ γρήγορα το θέμα των ε, ρυθμιστικών ε, τιμών αναφοράς και τις αρχές που τις διέπει σε σχέση με την ε, διαδικασία συλλογής, ιδιαίτερα από τις τρίτες χώρες, το άρθρο 1.1.24α γίνεται λόγος για τους ε, διαχειριστές που λαμβάνουν στοιχεία από τρίτους και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ε, τηρούνται οι αρχές εξωτερικής ανάθεσης που ορίζονται από το άρθρο 10. Για τους δείκτες αναφοράς όμως θα συνεργαστούμε με τους αποκοινού νομοθέτες και τους εμπλεκόμενους φορείς για το επίπεδο 1, έτσι ώστε εάν αλλάξει το επίπεδο 1, αν το αποτέλεσμα που είναι απότοκο του επίπεδου 1, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Τελικά σχόλια από την Καρολίν, την εισηγήτριά μας. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ τους ε, Σκιώδης και την Επιτροπή. Καλωσορίζω τα σχόλια του κυρίου Φερνάντες και της Επιτροπής και θα συνεργαστούμε εκ του σύνεγγης. Ε, σε σχέση με τους κρίσιμους δείκτες αναφοράς θα ήθελα να είμαι σίγουρη ότι δεν θα υπάρχουν κλειδονισμοί στην αγορά και θα παρακολουθήσουμε αυτό το θέμα εκ του σύνεγγυς τους επόμενους μήνες. Αυτά είναι τα σχόλιά μου σε αυτό το επίπεδο συζητήσεων. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι ολοκληρώνονται οι συζητήσεις και θα κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 10 για το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. So, hello everybody. We continue our meeting. Να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας, λέει ο Πρόεδρος, και καταρχάς να κάνω μια επιπλέον ανακοίνωση. Το αποτέλεσμα της κοινής, του κοινού τρογημερής διαλόγου σε ό,τι αφορά την ε, επανεκταστασία ΕΜΑ για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, λοιπόν, αρχή ε, που έλαβε χώρα 9 Ιουλίου του τρέχοντος έτους και οι συνομοθέτες ενέκριναν το αποτέλεσμα της τεχνικής συνάντησης της 10 Ιουνίου και η συμφωνία για τα υπόλοιπα ζητήματα, τα κρεμή ζητήματα σε ό,τι αφορά την έδρα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων δεν έχει ακόμα εξευρεθεί μεγάλη έκπληξη. Η Προεδρία λοιπόν θα ζητήσει νέα εντολή που θα επιτρέψει στους νομοθέτες να ολοκληρώσουν γρήγορα τις διαπραγματεύσεις με ειδική διαδικασία. Άρα πιστεύουμε και υπολογίζουμε στην Αυστριακή Προεδρία να επιλύσει το μεγάλο αυτό θέμα. Και τώρα να περάσουμε στο σημείο 4, 5 και 6 της μερισίας διαταξή μας, που είναι ο κανονισμός για την τροποποίηση κανονισμών που θεσπίζουν οι Ευρωπαϊκέ Εποπτικές Αρχές και κανονισμών σχετικά με τις χρηματοοικονομικές αγοράς. 1093 του 2010, 1094 του 2010, 1095 του 2010, 345 του 2013, 346 του 2013, 600 του 2014, 2000, 760 το 2015, 11 το 2016 και 112 του 2017 για την ε, μεταρρύθμιση της ΕΣΑ λοιπόν μιλάμε. Και χαίρομαι που είναι εδώ και οι δύο συνεισηγητές. Ελπίζω όλοι σας ε, να διαβάσατε χθε το βράδυ τα email σας που λάβαμε τα πρώτα σχέδια. Σήμερα θα ακούσουμε την παρουσίαση και να δώσω το λόγο στους συνεισηγητές. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπούρχαρτ Πάλτσα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Α, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο Πρόεδρος τον ανέφερε ήδη. Το σχέδιο έκθεσης ε, το λάβαμε χθες ε, το βράδυ. Το λάβατε μάλλον το χθες το βράδυ και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτή. Δεν σκοπεύαμε να υποβάλουμε το σχέδιο έκθεσης ε, τόσο καθυστερημένα ως αλλά μέχρι την τελευταία στιγμή πραγματικά κάναμε διαπραγματεύσεις όλοι οι συνεισηγητές. Υποβάλαμε λοιπόν τις εκτάσεις πλέον και θεωρώ ότι κάναμε ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω διαδικασία σε ό,τι αφορά τις προτάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανοίγουν την ενθεώρηση 12 ε, νομοθετικών προτάσεων ε, πάρα πολλέ σελίδε, εκατοντάδε. Μετά από εννέα μήνε εργασία, λοιπόν, θεωρώ ότι έχουμε σημειώσει μια κάποια πρόοδο. Λίγο παραπάνω από ότι το Συμβούλιο. Αυτό που κατέστη σαφέ ήταν ότι δεν ήταν δυνατόν να συμφωνήσουμε στο ίδιο βαθμό σε όλα τα θέματα. Παρά το γεγονό ότι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει γρήγορα να εξετάσουμε τα θέματα αυτά. Άρα, σε ποια σημεία συμφωνήσαμε καταρχάς, σε ό,τι αφορά την επεξεργασία της ΕΠΑ, ΑΙΟΠΑ και ΕΣΜΑ. Καταφέραμε να συμφωνήσουμε σε ό,τι αφορά την ενίσχυση τη αναλλαγικότητα, τη εργασία των Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτεία. Υπάρχει μια γενική ανάγκη για να υπάρχει αναλογικότητα στην ε, πρόταση. Και αυτό μπήκε και στον ε, εγχειρίδιο της ε, ΕΣΑ και της ΕΣΜΑ, της Ευρωπαϊκής Επιπτικής Αρχής. Αυτό λοιπόν θέλουμε να ληφθεί υπόψη στο μέλλον όλο και πιο πολύ. Θέλουμε επίση το Συμβούλιο Καταγγελίων να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως σώμα ελέγχου και θέλουμε να υπάρχουν πιο πολλές, ε, να εισακούγεται πολύ η φωνή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και όχι μόνο με την ε, πλειοψηφία δύο τρίτων, αλλά και ως μεμονωμένοι εκπρόσωποι της ομάδας. Κατά δεύτερον, συμφωνήσαμε σε ό,τι αφορά την ε, παροχή πρακτικών σε ό,τι αφορά τις συνεδριάσεις των σωμάτων λήψη αποφάσει. Αυτό θεωρώ ότι θα βελτιώσει τη λογοδοσία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και στα ό,τι αφορά το SSM και το SRB. Εδώ υπάρχει υστέρηση. Αυτό λοιπόν θέλουμε να το διορθώσουμε με την πρότασή μα. Γιατί οι Ευρωπαϊκέ Αποπτικέ Αρχέ έχουν ένα δημόσιο λειτουργήμα, τον δημοκρατικό έλεγχο. Και στη τελική ανάλυση θα πρέπει να είναι δημόσια τα πρακτικά αυτά. Τρίτο σημείο καταφέραμε να συμφωνήσουμε και για τη διευκρίνηση της εντολής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Αυτό η Επιτροπή μας το ζητά εδώ και πολύ καιρό. Το θεωρεί πολύ σημαντικό στοιχείο. Και στο σχέδιο έκθεσης αυτό αναφέρεται λοιπόν ε, η... ο περιορισμός των γνωμοδοτήσεων των ε, αρχών αυτών που συνδέονται με τη λόση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ό,τι αφορά επίσης ε, τον ορισμό των questions and answers, των έρωτα απαντήσεων. Αυτό τώρα ήταν ε, σε μια γκρίζα ζώνη. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι αυτέ οι ερωταπαντήσει δεν είναι δεσμευτικέ και ότι ενδεχομένω να υπάρξουν άλλε εθνικέ λύσει και ότι καταρχά θα πρέπει να ελέγχεται κατά πόσον μπορεί να δοθεί απάντηση από τι εθνικέ αρχέ. Επίση, συμφωνήσαμε ότι επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ένα καταμερισμό των κατευθυντηρίων γραμμών των υποπτικών αρχών στο μέλλον. Αν ζητούνται και απαιτούνται από, ευρωπαϊκές, ε, από ευρωπαϊκή νομοθεσία ε, η χάραξη τέτοιων κατευθυντηρίων γραμμών, τότε θα ακολουθείται ο κανόνα των δύο τρίτων πλειοψηφία. Αν οι κατευθυντήριε γραμμέ προκύπτουν από ίδια πρωτοβουλία των υποπτικών αρχών, τότε το όριο αυτό είναι πιο χαμηλό. Ε, κανονική, απλή πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο μπορούν να ζητήσουν αιτιολόγηση της χρηματοδότησης από τις Ευρωπαϊκές Επιπτικές Αρχές και μπορούν να ζητήσουν και επίσης αναπομπή και απόσυρση των κατευθυντήριων γράμμων αυτών από πλευρά των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Χαρών. Επίσης, ε, ενισχύσαμε τον ρόλο του Συμβουλίου Προσφυγών. και σε ό,τι αφορά τον πεδίο εφαρμογής το οποίο θέλαμε να το διευρύνουμε για να τηρηθεί η αναλογικότητα την οποία και ανέφερα προηγουμένω. Στη συνέχεια, οι συνεισηγητέ. Συμφώνησαν επίσης για μεγαλύτερη χρήση της διαδικασίας διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτές οι διαβουλεύσεις λοιπόν μπορούν να καταστούν ο κανόνας όταν μιλάμε για την χάραξη κατά των τρίγων γραμμών. Οι διαβουλεύσει λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ευρέω και θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη α, ποικιλομορφία σε ό,τι αφορά του παράγοντε τη αγορά που συμμετέχουν. Πέμπτο σημείο. Καταφέραμε να συμφωνήσουμε για την υψηλή ποιοτική αξίωση σε ό,τι αφορά τα αποσπασμένα άτομα στι ομάδε των εμπλεκομένων φορέων. Για τη συντελική ανάλυση θα λάβει όλο και πιο μεγάλη ευθύνη το σώμα αυτό. Άρα η ομάδα των εμπλεκομένων φορέων θα τοποθετείται και για τις γνωμοδοτήσεις και για τις ερωτοπαντήσεις. Έκτο σημείο επί το οποίο επίσης συμφωνήσαμε να έχει συναπόφαση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου. Εδώ τα τελευταία χρόνια Υπάρχουν ε, κάποιες ε, συνεπτικές, ε, συνεκτικές εξέλιξεις τα τελευταία χρόνια και θα θέλαμε λοιπόν να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά και το, την ισορροπία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πέμπτο σημείο, έβδομο σημείο, συγγνώμη. Συμφωνήσαμε και για την αξίωση να υπάρχει με καλύτερη υποπτική αρμοδιότητα σε διεθνέ επίπεδο και άρα θα πρέπει να υπάρχει συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο καλό συντονισμό. Και νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε πιο σημαντικά τη συζήτηση για την πλήρη συμμετοχή ω μέλη των Ευρωπαϊκών Υποπτικών Αρχών σε διεθνεί ε, συμβάσει. Εκ παραλίλου, οι αρμόδιοι φορεί των Ευρωπαϊκών επιπτικών Αρχών θα πρέπει να οργανωθούν με καλύτερο τρόπο και να ζητηθεί εντολή για το Εποπτικό Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του στου διεθνεί αυτού οργανισμού. Κατά ογδόν, Βελτίωση τη νομοθετική διαδικασία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον καθορισμό προτύπων για τα RTS και τα ITS. Και εδώ, λοιπόν, έχουμε να διδαχθούμε πολλά από το παρελθόν. Θα πρέπει να αυξήσουμε, λοιπόν, την ε, προβλεψιμότητα των μελλοντικών σχεδίων και να υποχρεώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει αναλόγως σε ό,τι αφορά αυτά τα quick fix, τις ε, βραχυπρόθεσμες αυτές τις προσαρμογές. Είχαμε πολλά στα τελευταία χρόνια. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν στο μέλλον θα θέλουμε να το περιορίσουμε. Πέραν από αυτό, στις εκθέσεις, στα σχέδια εκθέσεων, ζητάμε μεγαλύτερο ρεαλισμό σε ό,τι αφορά τα stress test, αυτές τις δοκιμές ε, αντοχής. Οι συνεισηγητές λοιπόν πιστεύουν ότι αυτές οι δοκιμές θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νομοθετικές ε, αξιώσεις, να έχουμε το βασικό σενάριο και το σενάριο μεγαλύτερου κινδύνου. Ένα το σημείο. Στοχευμένη προς προσανατολισμούς των ε, αναθεωρήσεων ζεύγους. Σε ό,τι αφορά δηλαδή το χτένισμα των πρακτικών αυτών εποπτείας. Και θα πρέπει να επιδιώξουμε την επίλυση προβλημάτων, όπως είναι για παράδειγμα η έλλειψη ανεξαρτησίας, αλλά και σε ό,τι αφορά την παραβίαση, για παράδειγμα, ευρωπαϊκών προδιαγραφών κατά 10 Δέκατο στοιχείο. Συμφωνήσαμε και για την ε, περιορισμό των ε, γραφειοκρατικών διαδικασιών σε ό,τι αφορά τις αντιπροσωπείες. Έλεγχος εξάντε του, της εξωτερικής ανάθεσης ε, των αρμοδιοτήτων. Αυτό θέλουμε να καταργηθεί. Εντέκατο σημείο. Προδιαγραφές για αιτήματα για παροχή δεδομένων από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Εδώ θέλουμε να απλοποιήσουμε το πολύ πολύπλοκο σύστημα το οποίο έχει καθιερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως να προτείνουμε και πρόστιμα. Να συνεχίσουν να υπάρχουν πρόστιμα σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι προδιαγραφές. Αν και ίσως να περιοριστούν τα πρόστιμα αυτά. 12 το στοιχείο. Συμφωνήσαμε για την ενίσχυση της χρηματοδοτικής διαδικασίας μέσω μιας ιστορική ελέγχου. 13ο. Ένα σημείο το οποίο με απασχολεί όλος ιδιαίτερος. απασχολει ολος ο Περιορισμό περιορισμος των άμεσων αρμοδιοτήτων της ΕΣΜΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών. Στον κανονισμό Γιουβέκα και ΟΙΖΕΦ και την ε, οδηγία Ιωσέφ ε, Έχουμε το θέμα αυτό. Όλα αυτά λοιπόν τα σημεία ήταν ε, σημεία στα οποία καταφέραμε να συμφωνήσουμε. Και τώρα να αναφέρω στο σχέδιο, να περάσω στο σχέδιο έκθεση, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Η και εγώ είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε μία συνάντηση του τη Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Και η εντύπωση που μα δόθηκε είναι ότι η διαχείριση ή διακυβέρνηση του Συμβουλίου αυτού θα πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά. Συζητήσαμε την δημιουργία ενός ε, ε, διευθυντή σε ό,τι αφορά τις θέσεις, ε, θέσεις του Διευθυντή για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό που θα επιτρέψει την καλύτερη λειτουργία του Συμβουλίου. Ωστόσο, δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα για την διατύπωση αυτή. Σε κάθε περίπτωση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, διευκρινίζουμε ότι θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό εκτός ε, του προπολογισμού της ΕΚΤ και ότι το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου θα πρέπει να επιμείνει πιο πολύ σε θέματα διαβούλευσης και θα πρέπει να αναπτύξει πιο πολλές τομεακές αρμοδιότητες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βγάλει, αν θέλετε, ε, το καπέλο της ε, τραπεζικής αρμοδιότητας και να κοιτάξει και άλλες ε, αρμοδιότητες και άλλους τομείς από τεχνικής άποψης. Από τα πολλά θετικά στοιχεία της εργασίας μου, της μας, θα ήθελα να αναφέρω και τα σημεία στα οποία δεν συμφωνώ. Είναι τα εξή. Δεν συμφωνήσαμε για το στρατηγικό σχέδιο επιτήρησης. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι σχέση δασκάλου-μαθητή. Πρέπει να αφήσουμε τις αποφάσεις στις εθνικές αρχές. Γιατί αυτές οι αρχές ε, πρέπει να ιδιολογήσουν τη χρήση πόρων και προσωπικού. Να μην ξεχνάμε ότι περισσότερη γραφειοκρατία δεν σημαίνει πάντα καλύτερη επιτήρηση. Γενικά, δεν συμφωνώ ότι πρέπει να αποδυναμώσουμε τις εθνικές ε, ελεγκτικές αρχές όπως προτείνει η Κομισιόν. Εγώ θεωρώ ότι έχουν γνώση, έχουν τεχνογνωσία και αυτή είναι και η γνώμη της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, στην ε, αναθεώρηση των εποπτικών αρχών. Επίσης, δεν συμφωνήσαμε για ουσιώδη θέματα της διακυβέρνησης. Στα σχέδια εκθέσεων ασχοληθήκαμε και με το ε, Διαχειριστικό Συμβούλιο και με το Εκτελεστικό Συμβούλιο που θεωρούμε ότι μπορούν να είναι ισότιμα. Για τη χρηματοδότηση θέλουμε να διατηρήσουμε το σύστημα και ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτήσεων αλλά δεν συμφωνήσαμε σε τι βαθμό οι ιδιωτικέ χρηματοδοτήσεις πρέπει να ε, συμβάλλουν στα οικονομικά των ε, οργανισμών επιτήρησης. Επίσης, δεν συμφωνήσαμε για ορισμένες από τις ε, άμεσες αρμοδιότητες των εποπτικών αρχών. Εγώ είμαι κάπως πιο περιοριστικός από την ε, συνεισηγήτριά μου. Θέλω να ληφθεί περισσότερο υπόψη ότι ορισμένα νομοθετήματα, όπως για τις τιμές αναφοράς ή για το εγχειρίδιο, έχουν μόλις ε, εγκριθεί. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει πάλι να τις αλλάξουμε τόσο σύντομα μετά την έγκρισή τους. Και δεν συμφωνήσαμε επίσης για το θέμα της διακυβέρνησης του CCP και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ξέρουμε ότι δεν ε, έχουν ολοκληρωθεί και άλλα νομοθετήματα. Οπότε είναι δύσκολο να ολοκληρώσουμε την αναθεώρηση των υποπτικών αρχών. Λοιπόν, ποιο είναι το προσωρινό μου συμπέρασμα. Είναι σαφές ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας ως Επιτροπή τους επόμενους μήνες. Τα σχέδια εκθέσεων, κατά τη γνώμη μου, συνολικά εκφράζουν ε, τη δυσαρέσκειά μας με τις προτάσεις της Κομισιόν. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Το μεγάλο θέμα της διακυβέρνησης και της χρηματοδότησης θα επιληθούν δύσκολα. Ακόμη και αν εργαστούμε μαζί. Γιατί θέλουμε να δούμε πώς θα καθοριστεί ο ρόλος και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής και των Εθνικών ε, Εποπτικών Αρχών. Θέλουμε να συνεργάζονται, όχι να αντιπαρατίθεται. Κατά τη γνώμη μου, όπω είναι τώρα οι προτάσει Κομισιόν δεν βοηθούν προ αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό πρέπει να βελτιωθούν. Αυτό θα επιχειρήσω να κάνω. Και έχω εμπιστοσύνη ότι και οι συνάδελφοί μου του ΕΛΚ εδώ στην Επιτροπή θα συνεχίσουν να εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να τονίσω επ' ευκαιρία για να ευχαριστήσω τη Γραμματεία της Επιτροπής και ιδιαίτερα τις δύο συνεργάτριες για την καταπληκτική βοήθεια που μας δώσανε και θέλω να ευχαριστήσω και την συνεισηγήτριά μου για την εργασία που δεν ήταν πάντα απλή αλλά δεν περιμέναμε ότι θα ήταν και τέλος τονίζω ότι εργαστήκαμε σκληρά τους τελευταίους μήνες και αυτό δεν έχει να κάνει αλλά μάλλον καλύτερα ότι η εργασία αυτή θα μας βοηθήσει όπως μας βοήθησε για τη διατύπωση των ε, εκθέσεων και στη διατύπωση των τροπολογιών που ενδεχομένως θα κάνουμε τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάλτς. Να δώσω το λόγο στην συνεισηγήτριά σας, κυρία Περβάνος Μπερές. Ευχαριστώ. Ε, ίσως πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη που μας πήρε τόσο χρόνο. Όπως έλεγε ο Φασμάν Μιτράν, πρέπει να δώσουμε χρόνο στο χρόνο. Και ήταν αναγκαίο για το θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα, κάθε συνεισηγητής ε, έπρεπε να κατανοήσει, να χωνέψει τα τόσο μακροσκελή κείμενα. Και ίσως κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε καλά όλο αυτό το χρόνο για αυτό το αποτέλεσμα το χρειαστήκατε. Αλλά εδώ καταλήξαμε. Όπως είπε και ο συνάδελφος Μπάλτς, ο συνσηγητής μου, κάτι που είπε ως κατάληξη, εγώ θα το πω σε εισαγωγή. η συνεργασία με τους συναδέλφους ε, του ΕΛΚ και της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, του, της Τσέντεου της Γερμανίας, είναι θετική. Γιατί ο καθένας εμένει επί των ε, θέσεών του και παρόλα αυτά καταλήγουμε σε, προσπαθούμε τουλάχιστον να καταλήξουμε σε κοινή θέση. Ξέρετε, νομίζω ότι αποδείχθηκε για το θέμα αυτό ότι το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Αν θέλουμε κάπου να καταλήξουμε, αυτά που σας υποβάλλουμε σήμερα, ίσως είναι απλώς ε, περιορισμός των ζημιών, αλλά ίσως μπορεί να χαρακτηριστεί και σημείο ισορροπίας. Οπότε ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Πριν μπω στις λεπτομέρειες, με το ίδιο πνεύμα με τον συνεισηγητή μου, αναφέροντας τα σημεία συμφωνίας και διαφωνίας, μια τελευταία προκαταρκτική παρατήρηση. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του πακέτου. Το συζητήσαμε όταν ε, παρουσιάστηκε το εγγραφό Αλλά αν δούμε τους στόχους ε, θα έχουμε μια καλύτερη περιχαράκωση των σημείων συμφωνίας και διαφωνίας. Ξέρετε ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι υποβολής αυτού του πακέτου. Θέλω να τονίσω έναν μόνο οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι πολύ διαφορετικές. Άρα υπάρχει ανάγκη να καθορίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τους όρους ισότιμης συνεργασίας για να σεβαστούμε και την ε, αναλογικότητα σίγουρα αλλά για να προωθήσουμε και την ε, ανάπτυξη μιας κοινή αντιμετώπισης. Φυσικά δεν θα ελέγχουμε ε, κάθε λεπτομέρεια της λειτουργίας των εθνικών αρχών, αλλά θα πρέπει να μην υπάρχουν κενά στην ε, προσέγγισή μας. Πρέπει να τα κλείσουμε. Πού συμφωνούμε. Επιβεβαιώνω αυτά που είπε ο συνάδελφος Μπάλτς, αλλά θα πάω και λίγο, πια, λίγο παραπέρα. Γιατί δεν τα ανέφερε όλα και θεωρώ ότι αξίζει να αναφερθούν σε αυτή τη φάση της συζήτησης. Εξετάζοντας την ουσία των προτάσεων της Επιτροπής. Όλα τα θέματα λογοδοσίας, ρόλος του Κοινοβουλίου, η προσθήκη κάποιων σημείων που δεν τα έχει αναφέρει καθόλου η Κομισιόν, τα άρθρα 10 έως 16, για τα RTS, τα STS, και με συγχωρείτε εάν δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ, είναι η νομοθεσία επίπεδου 2 και 3. Δεν είχε πει τίποτα κομισιόν για αυτά. Εμείς την συμπληρώσαμε αυτή την, ε, αυτό το τμήμα του κειμένου με βάση και την πείρα του Κοινοβουλίου. Όπως απεδείχθηκε στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε για διάφορους δείκτες. Εδώ ε, δώσαμε περισσότερες δυνατότητες στη διαβούλευση, και καθορίσαμε πιο συγκεκριμένα και πιο καθαρά το ρόλο των έρωτα απαντήσεων που είναι τελικά δυνατότητες που τις χρησιμοποιούν ιδιαίτερα οι, οι εποπτικές αρχές αλλά ξέρουμε ότι κάποια φορά οι εθνικές αρχές τις κάνουν σχεδόν δεσμευτικές γιατί με χαρά καλύπτονται πίσω τους για να μην χρειάζεται να κάνουν σωστά τη δουλειά τους ποιες είναι οι πραγματικές αρμοδιότητες που προβλέπει η πρόταση της Επιτροπής. Να τις αναφέρω με τη σειρά. Για το στρατηγικό σχέδιο. Το ανέφερε ο Μπούρκαρτ Μπάλτς, είπε ότι είναι σημείο διαφωνίας μεταξύ μας. Αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει δυνατότητα για, ένα, για στρατηγικά σχέδια που να θεωρούνται σχέδια της Ένωσης, που δεν αντιτίθενται με τα στρατηγικά σχέδια των εθνικών αρχών. Με την απέτηση βέβαια ότι θα λαμβάνεται υπόψη ο διαφορετικός τρόπος λειτουργίας, το διαφορετικό business model στον τραπεζικό, ασφαλιστικό ή τον τομέα των αγορών. Ο ρόλος των επιθεωρήσεων από των εθνικών αρχών. Συμφωνήσαμε για ένα κατά τη γνώμη μου ισορροπημένο και πρωτότυπο τρόπο που δεν ε, ε συμπεριλαμβάνει τον όρο αξιολόγηση ομοτήμων, peer review. Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να ε, αλλάξει η νοοτροπία με βάση τα διδάγματα από το παρελθόν. Αν μια εθνική υποπτική αρχή δεν κάνει σωστά τη δουλειά της, κάποιος πρέπει να διορθώσει την κατάσταση. Και ο καλύτερος τρόπος να το κάνουμε είναι να γίνει ένας ε, έλεγχος, μια επιθεώρηση με ένα από τα υψηλά ιστάμενα μέλη της ε, αρμόδιας Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής που θα έχει την ευθύνη για πέντε εθνικές εποπτικές αρχές που να κάνει την επιθεώρηση και αν χρειάζεται να δημοσιεύσει και την έκθεση για τα θέματα των εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια διάκριση για αυτές που είναι εντός και εκτός της Ένωσης. Είπαμε επίσης ότι πρέπει να ενημερώνεται τακτικά το Κοινοβούλιο για όλες τις αρμοδιότητες αυτές της Κομισιόν. Στο άρθρο 35 για τη συλλογή πληροφοριών αναγνωρίζω ότι απλουστεύσαμε κατά πολύ την πρόταση της Επιτροπής που ήταν τρομερά φιλόδοξη ίσως λίγο υπερβολικά σε αυτή τη φάση ε, εξέλιξης των λειτουργιών των εποπτικών αρχών και νομίζω ότι αυτό που τελικά συμπεριλάβαμε στην, στην ε, έκθεσή μας είναι η βέλτιστη λύση. Για τις ομάδες ε, ενδιαφερομένων ή εμπλεκομένων φορέων, stakeholder group, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει σωστή κατανομή μεταξύ των δύο ομάδων, δηλαδή συγκεκριμένα 13 για, τις ε, μεγάλες, ε, για τους μεγάλους φορείς και 12 για τις μικρότερες ομάδες και 4 συμπειρογνώμονες. Για τη διακυβέρνηση, ναι, διαφωνούμε. Αλλά σε ένα σημείο συμφωνούμε απόλυτα, και νομίζω ότι είναι μια πρωτότυπη πρόταση που θα πρέπει να εφαρμοστεί. Να υπάρχει μια επιτροπή επιλογής για να να εμβαθύνουμε την εμπλοκή μας στην αγορά, να έχουμε δηλαδή κάποια άτομα που να μπορούν να βοηθήσουν να καθοδηγήσουν αυτές τις αρχές. Τέλος. Ποιος θα κάθεται γύρω από το τραπέζι. Όταν οι οργανισμοί αυτοί εγκρίνουν ε, νομοθετήματα επίπεδου 2, σήμερα συμμετέχουν οι εθνικές εποπτικές αρχές. Αλλά οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί είναι και ρυθμιστικοί και εποπτικοί οργανισμοί. Και γι' αυτό συμφωνήσαμε ότι όταν ασκούν ε, ρυθμιστικές αρμοδιότητες, οι εθνικοί εκπρόσωποι δεν θα είναι οι εποπτικές αρχές, αλλά οι ρυθμιστικές αρχές, αυτές που δρούν σε επίπεδο 1, δηλαδή τα Υπουργεία Οικονομικών. Αυτά ε, για την προσπάθεια που θεωρώ ότι είναι και σημαντική και πρωτότυπη σε σχέση με την πρόταση τη Επιτροπή να δημιουργήσουμε μια νέα νοοτροπία που νομίζω θα σε ενδιαφέρει. Όπω ε, έκανε και ο Μπουρκρατ Μπάλτ, να αναφέρω σύντομα τα σημεία επί των οποίων ε, είτε σε αυτή τη φάση δεν έχουμε ακόμη συμφωνήσει είτε θα μπορούσαν να εξεταστούν και άλλες προτάσεις για τις ίδιες τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, όπως είπε και ο Μπουρκαρτ Μπάλτς, διαφωνούμε για τη διακυβέρνηση. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση της Επιτροπής. Με όλες τις, τις επιπτώσεις. Και για την ΕΣΜΑ να υπάρχει δυνατότητα η συμφωνία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο μας να ληφθεί υπόψη. Για το ρόλο δηλαδή της ΕΣΜΑ στην επιτήρηση των οργανισμών αποζημίωσης. Δεν συμφωνήσαμε όσον αφορά την ενίσχυση της προστασίας των ε, καταναλωτών με μια ευρεία ε, προσπάθεια ορισμού του τι σημαίνει καταναλωτής ε, για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει να είναι μέσα στην λειτουργία των και τη δραστηριότητα των υποπτικών οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα θέματα για την ΕΣΜΑ τώρα. Είπαμε ότι θέλουμε αυτό το προσπέκτους ε, να το κρατήσουμε, τον ορισμό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εγώ θα ήθελα να την κάνω πιο λειτουργική. Θα, θα ήθελα να κάνω πιο λειτουργικό αυτόν τον ορισμό. Προτείνω τροπολογίε ούτω ώστε η ΕΣΜΑ να συμπεριλαμβάνει και τα CCP και τα CDS και τα trade venue. όπως ακριβώς αναφέρθηκε κατά την αλλαγή απόψεων όταν υποβάλαμε το έγγραφο εργασίας. Για την ΕΙΟΠΑ, να ενισχύσουμε το ρόλο της προτώνω, προτείνω για τον έλεγχο των εσωτερικών προτύπων και να συμπεριλάβουμε τα απορίσματα που θα προκύψουν από τη συζήτηση για τα προϊόντα ΠΕΠ, τα προϊόντα συντάξεων, όπου η Επιτροπή δίνει κάποια εξουσιοδότηση στην ΕΙΟΠΑ που και εμείς ε, πιστεύω ότι θα συμφωνούμε μαζί της. Και τέλος, θα κάνουμε μια πρόταση για να ενισχυθεί ο ρόλος των ε, συλλογικών οργάνων επιτηρητών για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, που είναι πολύ λεπτό θέμα για τις ασφαλίσεις στον ασφαλιστικό τομέα, αλλά μπορεί να αφορά και τους δύο άλλους ε, θεσμούς. Τις δύο άλλες αρχές. Νομίζω ότι από αυτού θα μπορούσαμε να συνυποβάλουμε τροπολογίες. Σίγουρα και μακρηγόρησα και δεν ε, εξήγησα αρκετά κάποια σημεία, αλλά νομίζω ότι έτσι έχετε μια επισκόπηση της προόδου των διαπραγματεύσεών μας και του σημείου προόδου της έκθεσης. Λυπάμαι που δεν ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις μας ο Μπούρκαρτ Μπάλτς και εγώ και χαίρομαι που θα συνεργαστώ με όλους τους κοιόδης και με τον διάδοχο του Μπούρκαρτ Μπάλτς κατά το τελευταίο τμήμα της έκθεσης, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα η Σκιώδης, δεν υπάρχει κανείς από το ECR. Φιλελεύθερη, ο Βολφ Κλίνς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τους ε, δύο συνεισηγητές για την έκθεση αυτή. Τώρα δεν ξέρω να χαρώ που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την έκθεση πριν από τις θερινές διακοπές, γιατί προφανώς και είναι ενδιαφέρουσα η έκθεση, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολη και είναι και δύσκολο να τη διαβάσω το καλοκαίρι. Δεν είχα χρόνο να μελετήσω την έκθεση, το σχέδιο έκθεσης από χθε το βράδυ. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα κάνω οριστικά σχόλια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτά που έχετε ήδη ε, υποβάλει και σε ό,τι αφορά τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να αναφέρω ένα από του τρει τομεί ε, σε ό,τι αφορά την εντολή, την διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση. Σε ό,τι αφορά την εντολή. Όλοι ξέρουμε ότι η κρίση του 2008 ήταν ε, τέτοια έκταση. Μεταξύ άλλων, ακριβώς επειδή στην Ευρώπη είχαμε διαφορετικέ αντιλήψεις, διαφορετικές νοοτροπίες και διαφορετικό βαθμό αποτελεσματικότητας. Γι' αυτό λοιπόν και τότε και σήμερα συμφωνήσαμε για τη διατησία σε ό,τι αφορά τα θέματα ε, ρυθμισής και γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να υπάρξει μεγαλύτερη σύγκληση. Αυτός είναι ένας στόχος ο οποίος μας ενώνει, θεωρώ, και γι' αυτό καλό είναι και σωστό είναι όλα αυτά που συνέβησαν και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υπέβαλε μία πρόταση. Τώρα, η ακρόαση που είχαμε εδώ στην Επιτροπή μας με τους εκπροσώπους των εθνικών υπηρεσιών αλλά και με άλλους φορείς που εδώ και χρόνια ασχολούνται με το θέμα της ευρωπαϊκής εποπτείας κατέδειξε ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση απόψεων σε ό,τι αφορά αυτά που πιστεύουν οι ευρωπαϊκές εθνικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι αυτό μας παρουσίασαν και ως συμπέρασμα και οι συνεισηγητές. Άρα, ε, μια τέτοια αλλαγή νοοτροπίας δεν μπορεί να επιτευχθεί σε μια νυχτά, όπως προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να επιδιώξουμε σαφή πρόοδο, χωρίς ωστόσο να αμφισβητήσουμε την ίδια την εργασία και να αποδυναμώσουμε την ίδια την εργασία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, γιατί σίγουρα αυτό θα ήταν αντιπαραγωγικό. Γιατί αυτή η τελική ανάλυση είναι αυτοί που έχουν και την εμπειρία και την τεχνογνωσία. Δυστυχώ δεν είναι ε, εξίσου αποτελεσματικές όλες οι εθνικές αρχές. Γιατί κάποιες ε, ε, εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν ε, δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας και άλλες δυστυχώς απέχουν παρασάγκας. Και έτσι και πιο πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζουν και πιο πολύ χρόνο χρειάζονται για να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο εποπτείας. Σε ό,τι αφορά την, το, την εντολή και τις αρμοδιότητες. Εδώ θεωρώ ότι κάποια πράγματα είναι εντελώ ε, σίγουρα και μια αμφιλεγόμενα σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τι ε, εκτιμήσει από μοτίμου στο peer review. Θα πρέπει να φροντίσουμε ότι οι πιο αδύναμε εθνικέ αρχέ ε, θα μπορούν να διδαχθούν από τι πιο αποτελεσματικέ. Και αυτό προφανώ να μην γίνει με μια αντιμετώπιση δασκάλου και μαθητή, αλλά με έναν συναδελφικό τρόπο σε ό,τι αφορά τα στρατηγικά σχέδια τώρα και τη στρατηγική εποπτεία. Και στο σημείο αυτό είναι σαφές ότι για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια κάποια σύγκληση, θα πρέπει να υπάρχουν ενιαίοι στρατηγικοί στόχοι με κοινή διατύπωση και προκειμένου λοιπόν οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να παίξουν ένα ρόλο συντονιστή στο πλαίσιο αυτό και αυτό θεωρώ ότι είναι πέρα από κάθε αμφιβολία. Οι πιο πολλές αλλαγέ πιστεύω θα γίνουν ε, στην ΕΣΜΑ. Στην ΕΜΠΑ και στην ΑΙΟΠΑ θα γίνουν κάποιες αλλαγέ, αλλά θεωρώ ότι στην ΕΣΜΑ θα γίνουν πιο πολλές αλλαγέ, γιατί στα ΡΕΠΟΣ είναι πολύ αποτελεσματική και σε ό,τι αφορά τους οργανισμού επιστρεπτική ικανότητα, ε, και θα λάβει λοιπόν ε, και άλλες αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά τις τιμές αναφοράς, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, σε ό,τι αφορά το prospect είμαι λίγο πιο διστακτικό από ό,τι υπερβάνωσαν από την αλήθεια, γιατί γνωρίζουμε από τον CEO τι έγινε σε ό,τι αφορά τις τελευταίες εισαγωγές στα χρηματιστήρια. Το θέμα των prospect λοιπόν επιλύθηκε μια χαρά σε εθνικό επίπεδο, δεν χρειάστηκε ευρωπαϊκή εποπτεία στη τελική ανάλυση. Αυτό ενδεχομένω να μην ισχύει σε όλε τι περιπτώσεις, αλλά σε γενικέ γραμμές θεωρούμε ότι η ΕΣΜΑ θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για όλα τα prospect. Ε, και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύσει. Σε ό,τι αφορά τη χορήγηση ελέγχου αντιστοιχία και για τρίτες χώρε εδώ θα πρέπει να είναι αρμόδιο πάντα η ΕΣΜΑ προκειμένου να μπορεί να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα η ΕΣΜΑ κατά πόσον οι όροι και οι συνθήκες εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τις οποίες χορηγήθηκε αυτή η έγκριση. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο. Αυτό είναι απαραίτητο και θεωρώ ότι είναι θετικό το ότι αναφέρεται. σε ό,τι αφορά τον ΕΙΟΠΑ. Η υπερβάνουσα θέλει να δώσει μεγαλύτερο ρόλο στην ΕΙΟΠΑ σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές ε, διεργασίες. Εδώ θα ήθελα να επιδείξουμε προσοχή γιατί τα σχόλια τα οποία έχω ακούσει ως τώρα είναι ότι η ΕΙΟΠΑ ως τώρα έχει και κάπως μονομερή προσέγγιση, υπερβολικά μονομερή. Γι' αυτό λοιπόν να σκεφτούμε τον ρόλο που θα έχει η ΕΟΠΑ και στο μέλλον. Και για άλλα ζητήματα σε ό,τι αφορά τα ΠΕΠ, για παράδειγμα. Επί της αρχής συμφωνώ, η ΕΙΟΠΑ, εφόσον ε, εισαγάγουμε ένα ευρωπαϊκό ε, προϊόν συντάξεων, να παίζει σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, να προσέξουμε, γιατί η ΕΙΟΠΑ συνολικά Είναι πάρα πολύ συντηρητική σε ό,τι αφορά τον θέμα των ασφαλιών και αυτό το προϊόν ΠΕΠ λοιπόν δεν θα θέλαμε να είναι ένα κλασικό προϊόν ασφάλειας. Θα θέλαμε να έχει μια τέτοια διάρθρωση προκειμένου να μπορέσει να παρέχεται και από άλλου ε, φορεί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Και εδώ θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε προσοχή. Κατά δεύτερον, για θέματα διακυβέρνηση. Πιστεύω ότι είναι πολύ φυσιολογικό και πολύ σωστό το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή στο σημείο αυτό, γιατί στην τελική ανάλυση το Επαπτικό Συμβούλιο, το οποίο έχει έχει όλες αυτές τις αρμοδιότητες είναι πάρα πολύ μεγάλο. 28 κυρίες και κύριοι που συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή λοιπόν και οι οποίοι προφανώς έχουν κατανόητα τα εθνικά συμφέροντα. Εδώ είναι απαραίτητο να έχουμε μία μικρή δομή, η οποία θα είναι ταχεία στην αντίδραση της σε ό,τι αφορά το εκτελεστικό συμβούλιο. Λοιπόν, αυτό χρειαζόμαστε, πιστεύω. Ο, η θα έχει λοιπόν την καθοριστική ψήφο σε περίπτωση ισοψηφία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρότεινα να μην έχουμε τέσσερα ε, μέλη στο εκτελεστικό αυτό, στην εκτελεστική επιτροπή, ή τρία ή πέντε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο, ο ή πρόεδρο να είναι αυτοί που θα έχουν ε, την καθοριστική ψήφο σε περίπτωση που χρειαστεί, λοιπόν, κάτι τέτοιο. Έγινε και μία δημόσια ακρόαση, λοιπόν, και πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και εξωτερικούς ε, παράγοντες στο πλαίσιο αυτό που δεν προέρχονται απαραίτητα από τις εθνικές επιπτικές αρχές. Ε. Ίσως να έχουν ε, τέτοια εμπειρία, αλλά να έχουν σίγουρα ένα διάλειμμα 2-3 ετών. Να έχουν όμως την τεχνογνωσία, χωρίς όμως να έχουν εθνικές, τα εθνικά συμφέροντα κατά νου απαραίτητα. η δομή εποπτείας είναι διαφορετική προφανώς στην ΕΣΜΑ από την ΕΣΜΑ και την ΑΙΟΠΑ. Γιατί έχουμε το θέμα του CCP. Δεν νομίζω ότι για το CCP χρειαζόμαστε ξεχωριστό, α, ξεχωριστές δομές. Αυτό θεωρώ ότι θα είναι υπερβολικό. Να υπάρχει κοινό συμβούλιο Πέντε ατόμων, για παράδειγμα, εκ των οποίων ίσω τα δύο 3 να ασχοληθούν με θέματα ΣΥΠΗ. Σε ό,τι αφορά του εμπλεκόμενου φορεί, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ, είναι να έχουμε και εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών, που να ασχολούνται όλο και πιο πολύ με τα θέματα τη προστασία του καταναλωτή. Γιατί αυτό έω τώρα δεν τονίζεται επαρκώ, πιστεύω να το επεκτείνουμε ως αρχή. Τρίτο θέμα. Χρηματοδότηση. Όποτε μιλάμε φυσικά για χρήματα, τα πράγματα δυσκολεύουν. Είπε ο Μπουρκάρτ ότι καταρχάς θα πρέπει ένα τμήμα, ένα 40% σε πρώτη φάση να προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπόλοιπο από τις εθνικές ε, ε αρχές εποπτείες. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή των ευρωπαϊκών αρχών, αλλά θα πρέπει να συμμετέχει και ο χρηματοπιστωτικό κλάδο στη τελική ανάλυση. Τώρα, σε τι ποσοστό ακριβώ, 60-40, 40-60, δεν ξέρω. Αυτό να το εξετάσουμε. Δεν μπορώ να σα πω την μαχική αναλογία. Αυτό που είναι σημαντικό, ωστόσο, είναι να βρούμε ένα μοντέλο το οποίο θα εξασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκέ εποπτικέ αρχέ θα εργάζονται με έναν αποτελεσματικό τρόπο ω προ το κόστο και να αναλάβουν ε, πλήρως τις ευθύνες τους. Και λογοδοσία και ευθύνη λοιπόν και ενώπιον ημών. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι, ότι δεν ε, σπαταλούνται χρήματα και πόρει. Άρα, συνολικά, θα έλεγα ότι είναι θετική εντύπωση μου το ότι καταφέραμε και κατάφεραν και οι συνεισηγητέ, ε, παρά τι διαφορέ ε, που είχαν ε, σε πρώτη φάση, να βρουν ένα συμβιβασμό σε πολλού τομεί. Νομίζω ότι στο Κοινοβούλιο θα καταφέρουμε συνολικά να βρούμε ένα συμβιβασμό ο οποίο θα υποστηριχθεί από όλε τι πλευρέ, λίγο πολύ. Είμαι πολύ διστακτικό ό,τι αφορά το Συμβούλιο, γιατί οι πρώτε αντιδράσει που ακούσαμε δεν είναι πολύ ευίωνες. Δεν θα είναι εύκολες οι διαπραγματεύσεις. Τώρα κατά πόσο θα καταφέρουμε πραγματικά μέσα στη θετία αυτή να κλείσουμε με επιτυχή τρόπο του τριμερείς διαλόγους δεν τολμώ να το προβλέψω στην παρούσα φάση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα παρακολουθήσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κλίντς. Ο Σβέν Γκίγκολτ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Βόλφ, ελπίζω, αν θες να διαβάσει κάτι καλύτερο, δώσου μου τη διεύθυνσή σου και θα σε εκπλήξει αυτό που θα σου στείλω. Γιατί θα ήταν κρίμα να έχεις να διαβάσει μόνο αυτή τη θαυμάσια έκθεση. Να έχεις να διαβάσει έξι εβδομάδες. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την εργασία των δύο συνεισηγητών, συνεισηγητριών. Είναι μια βάση επί της οποίας μπορούμε να εργαστούμε περιέχει πολύ ενδιαφέρουσες, συναρπαστικές ιδέες και προτάσεις που νομίζω ότι θα έχουν ευρεία πύχη στο Κοινοβούλιο, ιδιαίτερη ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου. Η προσπάθεια, οι εποπτικές αρχές να παίζουν ε, το ρόλο τους ε, στις, ε, στις διεθνείς στα διεθνή φόρουμ και με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει μια αποκοινοβουλευτικοποίηση ε, της προσπάθειας αυτής, συμφωνώ. Βεβαίως, καταλαβαίνω ότι αν έχουμε συνεισηγητές των δύο μεγάλων φιλοευρωπαϊκών ε, κομμάτων, ε, είναι λίγο απογοητευτικό να μην μπορούν να πούν ότι στηρίζουν την πρόταση της Επιτροπής ότι θέλει περισσότερη επιρροή των ευρωπαϊκών θεσμών στις εποπτικές αρχές. Αυτό το είπε και ο Κλίντς, αυτό είπαν και οι ακροάσεις, ότι το ευρωπαϊκό επίπεδο εκπροσωπείται λιγότερο από ότι τις ε, εθνικές αρχές. Φυσικά, θέλουμε να υπάρχει σχέση συνεργασίας. Θέλουμε να μην υπάρχει αντιπαράθεση εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου. Αλλά Νομίζω ότι όπως ε, είχε πει και το προηγούμενο κοινοβούλιο όταν ενέκρινε μια έκθεσή μου πριν από τόσο καιρό, πρέπει λοιπόν δεν αξιο... να τονίσουμε ότι δεν αξιοποιούνται πολλέ αρμοδιότητες των υποπτικών αρχών γιατί υπάρχουν προβλήματα και κενά στην διακυβέρνηση. Θα ήθελα λοιπόν ως Κοινοβούλιο να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα. Βεβαίω, θέλουμε ενίσχυση της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης της ε, ΕΣΑΣ και θέλουμε και εδώ υπερβαίνω και την πρόταση της Κομισιόν, θέλουμε να διαπραγματευτούμε με τα κράτη-μέλη, γιατί ξέρουμε τι θα προκύψει, θα πρέπει να διαπραγματευτούμε. Τώρα, στις προτάσεις για τη διακυβέρνηση υπάρχουν πολύ καλές και αναλυτικές προτάσεις. Να αναφερθώ στα εξή που δεν με πείθουν. Πρώτον, είναι πονηρό να λέμε ότι οι πρόεδροι των υποπτικών αρχών θα πρέπει να ε, ορίζονται για 8 χρόνια και καθ' όλη αυτή τη διάρκεια δεν θα μπορούν να ζητήσουν λογοδοσία ε, εμείς δεν θα μπορούμε να ζητήσουμε ε, λογοδοσία. Νομίζω ότι 2 επί 5 είναι καλύτερο, γιατί μετά από 5 χρόνια μπορούμε να κάνουμε μια νέα συζήτηση επί της αρχής. Και κάτι άλλο που δεν με βρίσκει σύμφωνο είναι αυτό που λέτε ότι, ότι μια επιτροπή των τριών θεσμικών οργάνων θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία προσφυγής. Και όπως λέει η 107 τροπολογία, αυτό λέει, και όχι να μην το σώμα μας συνολικά. Νομίζω ότι είναι μια ιδρυματοποίηση των δύο μεγάλων διαδικασιών. Βλέπω ότι όταν διαβάζει κανείς μια τέτοια έκθεση, σας παρακαλώ να μου διευκρινίσετε. Πεςτε μου, τι θέλετε να αλλάξει στη διαδικασία προσφυγής. Ε, συγγνώμη, η... ή διορισμού. Ε, πρέπει να τονίσω το εξή. Οι πρόεδροι των ε, εποπτικών αρχών ήταν πάντα υπόλογοι έναντι του Κοινοβουλίου. Και αυτήν την ε, λογοδοσία την υλοποιήσαμε με διάφορους τρόπους. Ε, δεν συμφωνούσαμε πάντα, αλλά την υλοποιήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Η, η κυρία Μπερές αναφέρθηκε σε δύο άλλα σημαντικά θέματα. Θα θέλαμε και ελπίζαμε ότι μετά την εργασία που κάναμε και που την τεκμηριώσαμε και με πολλές επιστημονικές μελέτες θα είχαμε και πορίσματα για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών για διάφορα θέματα επενδυτικών προϊόντων. Οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν κενά στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και υπάρχουν και παραβιάσεις του δικαίου για την εφαρμογή του δικαίου προστασίας των καταναλωτών. Και δεν έχει υπάρξει καμία διαδικασία από πλευρά των υποπτικών αρχών. Μόνο μια φορά για την ε, Βουλγαρία. Αλλά για πολύ σημαντικότερες περιπτώσεις ποτέ. Πρέπει λοιπόν οι υποπτικέ αρχές να ασχολούνται περισσότερο με την προστασία των καταναλωτών για να γίνει πραγματικότητα η ε, ένωση, η ένωση των κεφαλαίων Μόνο τότε θα υπάρξει μια πραγματική Ένωση κεφαλαίων Αγορών. Χρειάζεται ενίσχυση λοιπόν τη προστασία των καταναλωτών. Εδώ κάνατε κάποιε διαγραφέ ε, προτάσεων τη Κομισιόν. Μπορούμε να τι συζητήσουμε. Αλλά δεν βλέπω να ενισχύθηκε αρκετά αυτό που λέει για παράδειγμα το επιμελητήριο των επενδυτών και το επιμελητήριο των ε, καταναλωτών. Και κάτι ακόμη που ανέφερε και η και όπως συμφωνούμε, οι χρηματαγορές επίσης πρέπει να ασχοληθεί με την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να γίνουν περισσότερες επενδύσεις σε βιώσιμες μορφές ενέργειας. Δεν θέλουμε να υπάρξει νέα κρίση στις χρηματαγορές τώρα που επενδύουμε σε τέτοιες ε, βιώσιμες ε, προτάσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι στα καθήκοντα των ε, εποπτικών αρχών. Και αγαπητέ Μπάλτς, βεβαίως πρέπει να συμφωνήσουμε πώς θα νομοθετήσουμε σε κάθε τομέα, αλλά αυτό είναι κάτι κοινό. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν συμφωνήσατε από αυτού. Νομίζω ότι η βιωσιμότητα δεν θα έπρεπε να είναι επίμαχο θέμα, αλλά αυτονόητο θέμα μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει κάποιος από την ΚΟΕ, e, ούτε από την EFTD, ούτε από την ομάδα ENF. Catch ο κύριος Λάγκεν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ τους δύο συνεισηγητές και όχι, είχα άλλα πράγματα να κάνω αυτό το βράδυ, δεν διάβασα την έκθεση γιατί έχασα και το Βέλγιο, γιόρταζαν και οι Γάλλοι. Και τα ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν νομίζω ότι τα εξήγησαν καλά οι ομιλητέ για το μελλοντικό ρόλο των ε, Ευρωπαϊκών Υποπτικών Αρχών. Θα πρέπει να βασιστούμε και στις ε, εμπειρίες του παρελθόντος και ε, σε μία υπηρεσία έχουμε αρνητικές εμπειρίες στην ΑΙΟΠΑ και σε θέματα αναλογικότητα, αλλά και σε ό,τι αφορά τον ρόλο της ΑΙΟΠΑ για τις ε, κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες έχουμε θέματα. Και εδώ να ξεκινήσω λέγοντας το εξής, ε, ότι μετά την επανεκλογή του επικεφαλής του ΑΙΟΠΑ αμέλησε το Κοινοβούλιο. Στο παρελθόν τουλάχιστον ε, είχε κάποια διάθεση συνεργασίας. Γι' αυτό λοιπόν τα θέματα των κοινοβουλευτικών δικαιωμάτων μα εδώ, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί πολύ αμφιβάλλω κατά πόσον οι εθνικέ εποπτικέ αρχέ προωθούν την ευρωπαϊκή αυτή νοοτροπία. Και θα πρέπει να περάσουμε μια νέα ισορροπία. Η χρηματοδότηση εδώ και καιρό αποτελεί αμφιλεγόμενο και ακαντόδε σημείο. Εγώ επί της αρχής πιστεύω ότι συμφωνούμε σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της εθνικής ε, χρηματοδότησης, αλλά όχι να φτάσουμε στο σημείο να μην ε, μπορούμε να κληρώσουμε σημαντικά μέτρα σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την ε, εποπτεία των CCP. Αμφιβάλλω σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κύριος Κλίντσα. Θεωρώ ότι είναι νομοθετικές προτάσεις σε ό,τι αφορά την, το CCP είναι και σε ό,τι αφορά την δημιουργία ανάλογη ρυθμίση για το ΕΣΜΑ σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της αναλογικότητας. Είναι σαφές ότι η ΑΙΟΠΑ, επανέρχομαι στο σημείο αυτό, έχει πάρα πολύ σύνθετο και περίπλοκο σύστημα. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές λοιπόν έχουν την... δεν αξιοποίησαν τις δυνατότητες που υπήρχαν και η ΕΟΠΑ θέλει να έχει τη δυνατότητα. Έχει ποσοτικά υπερβολικά μεγάλο ο, συμπίλημα. Και όλα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα τακτικό πλαίσιο. Αυτό για να ορίσουμε και μόνο με σαφή τρόπο τις ε, εργασίες της ε, Στην έκθεση, η οποία είναι πάρα πολύ καλή λοιπόν, πιστεύω ότι εισαγάγεται με σωστό τρόπο και βελτιώνεται μάλιστα η αρχή τη αναλογικότητα. Καθώ και την ε, συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ποια μορφή θα συνεχιστεί. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια από τους συναδέλφους. Η Επιτροπή μόνο μας ακούει σήμερα. Πάντως ε, είστε πάντα ευπρόσδεκτοι να σχολιάσετε όποτε θέλετε. Δίνω το λόγο στους συνεισηγητές Burkhardt. Ευχαριστώ και θα είμαι σχετικά σύντομος να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις και να τονίσω οι ιδιαιτέρους αυτά που είπε ο συνάδελφος Κλίντς. Φυσικά βρισκόμαστε στο τέλος ενός ε, μεγάλου δρόμου, του δρόμου σύγκλησης. Αυτό είναι άλλωστε πιστεύω και ο στόχο των πιο πολλοπολιτικών ομάδων εδώ πέρα στην Επιτροπή μα. Ω εκ τούτου. Πιστεύω ότι αυτό ο γενικό και απότερο στόχο ε, δεν συζητιέται καν. Τώρα, αυτό που θα εξακολουθήσει σε κάθε περίπτωση να μας απασχολεί στο μέλλον είναι πραγματικά το πώς ε, οι αποκλήσεις μεταξύ των τριών ε, ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών και των εθνικών εποπτικών αρχών μπορούν να απαλληλθούν. Αυτό το είχα πει και πριν από κάποιε μήνε στην πρώτη συζήτηση ότι αυτό σίγουρα θα αποτελέσει ένα από τα βασικά καθήκοντα και μία από τι βασικέ εργασίε μα κατά την κατάρτιση τη έκταση αυτή. Και είναι πολύ θετικό, το είπα και εγώ ίδιο τον Τόνισε και ο συνάδελφο, το γεγονό ότι ασφαλώ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεδομένη και της διαφορετικής, ε, διαφορετικού επίπεδου τεχνογνωσίας και επαγγελματικότητα των διαφόρων εθνικών υπηρεσιών, θα πρέπει να υπάρξει μια νέα στήγοσταθμιση Προκειμένου ακόμα και οι μικρέ εποπτικέ αρχέ τελικά σε εθνικό επίπεδο να μάθουν και να διδαχθούν από τι άλλε που έχουν μεγαλύτερη τεχνογνωσία. Το θέμα διακυβέρνηση θα συνεχίσει να με απασχολεί και αυτό το παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον και στο μέλλον. Και όπως είπατε, όντως εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις το θέμα της χρηματοδότησης σε τελική ανάλυση πιστεύω ότι είναι επιλύσιμο. Βασικά το θέμα δεν είναι να αμφισβητήσουμε τη λειτουργία του αιτητού συστήματος. Υπάρχει μια σε τοποθέτηση και νομίζω ότι η Επιτροπή συμφωνεί ότι θα πρέπει να υπάρξει και στο μέλλον δημόσια χρηματοδότηση. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα ποσοστά. Να απαντήσω σε αυτά που είπε ο κύριος Σβέν Γκίγκολ. Εν συντομία και οι δύο πιστεύαμε ότι αυτή η οκταετή θετία ήταν καλή ιδέα. Και αυτό γιατί, γιατί όντω αυτό που είπε μόλις ο συνάδελφος Λάγκε ισχύει. Παρατηρούμε ότι κατά το πρώτο τμήμα της θητείας συχνά ε, δρούν με τρόπο πολύ φιλικό και κολακευτικό προς το Κοινοβούλιο και στο δεύτερο τμήμα της θετίας ε, δεν ισχύει αυτό ακριβώς έτσι για να το πω ουδέτερα. Άρα, μεγαλύτερη θετία θέλουμε, χωρίς επανεκλογή, αυτό και προτείνουμε και οι δύο μας. Ε, το τονίζω. Είμαστε πεπισμένοι ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν σκόπιμο. Γι' αυτό το βάλαμε άλλωστε και στα σχέδια έκθεσης. Και συνοψίζοντα, να πω ότι σίγουρα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσε οι συζητήσει συναρπαστικέ, αλλά νομίζω ότι πραγματικά οι δύο εκθέσει ε, αποτελούν μια καλή βάση για τι συζητήσει εδώ στην Επιτροπή. το τελευταίο θέμα το οποίο το ακούσαμε από τον συνάδελφο. Εγώ προσωπικά είμαι σχετικά βέβαιος ότι το Κοινοβουλίο στο σημείο αυτό θα σημειώσει αποτελέσματα και μάλιστα σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Θα περάσει σε ψηφοφορία στην Επιτροπή και είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Τώρα, κατά πόσον από την άλλη πλευρά, κατά πόσον ο νομοθέτη είναι εξίσου προετοιμασμένο, αυτό πρέπει να σας πω από δική μου πλευρά ότι δεν το γνωρίζω αγαπητέ Βόλφε, έχω τι αμφιβολίε μου. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι εμείς δεν πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα αυτό με προσήλωση και με μεγάλη φιλοδοξία, γιατί θέλουμε όσο πιο γρήγορα να, ολοκληρωθεί, να ολοκληρωθούν οι εκθέσεις στην Επιτροπή. Και με τον τρόπο αυτό προφανώς να σκίσουμε και μέσα πίεση στο Συμβούλιο. Θέλω να πω ευθέως ότι δυστυχώς πολύ αμφιβάλλω αν θα κινηθεί με αντίστοιχη ταχύτητα και επίπεδο φιλοδοξία και το, κοινοβούλιο, το Συμβούλιο. Συγγνώμη. έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ήταν παρόντες. Ξέρω ότι πολύ περισσότεροι θα διαβάσουν αυτή την έκθεση και θα συνεισφέρουν μέσω τροπολογιών θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις εγκαρσίου τύπου σε σχέση με την αρχική μας παρουσίαση. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τους οργανισμούς σε σχέση με μελλοντικά καθήκοντα που θα τους αναθέσουμε και σε σχέση με τις παρούσες αρμοδιότητές τους, γιατί διαφορετικά μπορούμε να πούμε οι οργανισμοί δεν μπορούν να κάνουν το τάδε ή το δίνα, αλλά θα πρέπει να ε, δεχτούμε ότι μπαίνουμε σε μία δυναμική πορεία. Ο Σβέν Γκίγκολτ ε, μίλησε ακριβώς για αυτή τη διελκυστίνδα που γίνεται μεταξύ όλων, δηλαδή τραβάν από εδώ, τραβάν από εκεί και κανείς δεν κινείται στο τέλος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κάτι ως προς τη διακυβέρνηση και τους οργανισμούς έτσι ώστε οι οργανισμοί που προϋπάρχουν και αυτοί που θα προκύψουν να μπορέσουν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Γιατί διαφορετικά δημιουργούμε αυταπάτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι το οποίο δεν είναι καλό ούτε για το Κοινοβούλιο ούτε για την Ευρώπη. Σε αυτό το θέμα της διακυβέρνησης κατανοώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε διαβλούς επικοινωνίας με τις διάφορες ομάδες. Τώρα, ε, κάτι το οποίο δεν αναφέραμε στην αρχική πρόταση θα ήθελα να προσθέσω, δηλαδή να προσθέσω δύο ή τρία στοιχεία. Σε κάθε κείμενα ε, υπάρχει ε, ένα στοιχείο προειδοποίησης και αυτό σε όλα τα κείμενα, γιατί υπάρχει και ο απόρριτος χαρακτήρας, η εχεμήθεια, γι' αυτό θα πρέπει να αντιλήσουμε από τα διδάγματα του παρελθόντος ως προς τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Δεν λέω ότι σήμερα ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα προειδοποίησης κατά της λειτουργίας των οργανισμών αλλά ένα γενικότερο σύστημα προειδοποίησης. Σε σχέση τώρα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, θα πρέπει να πω ότι η πρόταση της Επιτροπής ε, για να κερδίσει μία θέση στο Συμβούλιο, το οποίο έχει ευρύτατες αρμοδιότητες και ένα πολύ μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, ότι θα πρέπει δηλαδή να συμμετάσχει και ο οργανισμός ε, εξυγίανσης τη στιγμή που δεν υπάρχει πια το Επιστημονικό Συμβούλιο, θεωρούμε και είμαστε πεπισμένοι ότι η Επιστημονική Επιτροπή ε, δίνει μία ε, δυναμική πορεία στο Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, κάτι το οποίο χρειάζεται. Μετά την ε, επίσκεψη του Μάριο Ντράγκη θεωρούμε ότι με βάση τα θέματα που μας απασχολούν θα πρέπει να συμμετέχει σε τακτά χρονικά ε, διαστήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Κλίντς, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει πραγματικά να διατηρήσουμε το ρόλο όλων των ε, οντοτήτων αυτών και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μία πορεία προς τα πάνω. Ως προς το χρονοδιάγραμμα, συμμερίζαμε αυτά που είπε ο Μπούρχαρτ Βάλς. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με το χρονοδιάγραμμα του Συμβουλίου, αλλά αν μπορούμε να αποστείλουμε ένα μήνυμα προς το Συμβούλιο, είναι να έχει παραδειγματικό ρόλο σε σχέση με την έκθεσή μας και να αποδείξει έμπρακτα την ε, διάθεσή του για βελτίωση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των οργανισμών. Υπήρχε η αρχική πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με τη διαβούλευση που έγινε πιο ρεαλιστική και νομίζω ότι έμπρακτα μπορούμε να φέρουμε εις πέρα σε αυτή την πρόταση. Ο Σβέν ε, Γκίγκολτ μίλησε για την έκθεσή του, την έκθεση του 2014. Έχει ενσωματωθεί στο σκεπτικό μας και ως προς το διορισμό των προέδρων των ΕΖΑ υπήρχε η αρχική πρόταση της οκταετίας ο Σβέν Γκίγκολτ λέει ότι εάν ε, δεν γίνει αναθεώρηση στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή επαναδιορισμός, τότε αποδυναμωνόμαστε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω όμως ότι όταν γίνεται επαναδιορισμός τότε αποδυναμώνονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των οργανισμών. Το είδαμε αυτό έμπρακτα. Δηλαδή όταν ε, γίνεται επαναδιορισμός ή νέοι διορισμοί, τότε αποδυναμώνεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό σε σχέση με την Επιτροπή επιλογής. Ε, νομίζω ότι ο Σβέν θα ξαναδιαβάσει το έγγραφό μας γιατί κρατάμε την διαδικασία διορισμών ως έχει και την βελτιώνουμε με αυτή την Επιτροπή Επιλογής ε, Υποψηφίων. Θα υπάρχουν έξι μέλη, δύο από το Κοινοβούλιο, δύο από το Συμβούλιο και δύο από την Επίτροπη έτσι ώστε στην ουσία να κάνουν μία βολιδοσκόπηση της κατάστασης. Γιατί όταν έγιναν οι πρώτοι διορισμοί από την Κομισιόν των ΕΖΑ, η Επιτροπή επέλεγε αυτούς που είχαν τολμήσει να υποβάλουν υποψηφιότητα. Είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το θέμα, γιατί πολλοί δεν θέλουν να εκτεθούν, ε, φοβούνται για την ιστεροφημία τους και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να υποβάλουμε προτάσεις που μπορούν να ενταχθούν στην τακτική διαδικασία, όπως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών θα υποβάλω τροπολογίες και ο κύριος Μπάλτς ε, δέχτηκε τις ε, προτάσεις μου, ίσως κάπως καθυστερημένα, για να ενισχύσουμε το ρόλο του Διευθυντηρίου Εποπτών. Αυτές, αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές τη στιγμή που οι ρυθμιστικές αρχές δεν μπορούν να δουλέψουν καλά ως προς τον κύριο ε, Λάγκεν για την αναλογικότητα και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ ε, καλή βάση εργασίας και θα ήθελα να πω το χρονοδιάγραμμά μας είναι επιτακτικό πρέπει να τηρηθεί. Οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις διαπραγματεύσεις και θα ήθελα να πω ότι έχουμε ορισμένα τεχνικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίζουν γιατί το σύστημα θα ε, ανοίξει τέλη Ιουλίου αρχές Αυγούστου για τις τροπολογίες τη στιγμή που θα έχουμε και τη διάθεση της μετάφρασης. Θα σας πούμε πότε θα ανοίξει αυτό το μέσο 84am και ελπίζουμε μέχρι τα τέλη Αυγούστου, 30 Αυγούστου να έχουν υποβληθεί οι τροπολογίες. Έχουν έχουμε την Τρίτη, Τετάρτη και την Πέμπτη συνεδρίαση της ΕΚΟΝ. Τέλη του Αυγούστου. Βολφ, λυπάμαι, οι εισηγητές έχουν τον τελευταίο λόγο. Ποια είναι η πρόταση. Και αυτό είναι δικαίωμα των εισηγητών. Αν και συμφωνώ ότι θα πρέπει να κλείσει το ζήτημα το συντομότερο, θα ήθελα να παρατείνουμε την υποβολή τροπολογιών κατά μία εβδομάδα. Στις 5 Σεπτεμβρίου προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Κάτι τέτοιο. Επτά Σεπτεμβρίου για τις τροπολογίες. Ε, στις 5 τι λένε οι εισηγητές. Γιατί δεν θα είναι οι μεταφράσεις έτοιμες. Γιατί τώρα... Ναι, η έκθεση είναι στα αγγλικά, αλλά εκτός μικροφώνου παρατηρήσεις. Ναι, ο καθένας μπορεί να υποβάλει τροπολογίες στη μητρική του γλώσσα, αυτό είναι δικαίωμα. Θα λάβετε ε, ένα μήνυμα για το πότε ανοίγει αυτό το μέσο, ATM4M, και νομίζω ότι μέχρι τις 30 ε, Αυγούστου στις 12 ε, το μεσημέρι θα πρέπει να λάβετε γνώση αυτού του μέσου. Έχει γίνεται και Έχουμε και επιτροπή εκείνη τη βδομάδα και οι εισηγητές θέλουν να τηρήσουν την προθεσμία. γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει μόνο η θέση των συντονιστών, αλλά των εισηγητών, η οποία προέχει. Είναι πολύ δύσκολο να το κρίνω. 30 Αυγούστου στις 12 και στις, ε, την 1η Οκτωβρίου το, στο Στρασβούργο θα εξετάσουμε τις τροπολογίες, τη Δευτέρα το βράδυ του Στρασβούργου και στις 5 ε, Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε στην ΕΚΟΝ και εάν επιτευχθεί συμφωνία μετά τον τριμερή στις 12 Νοεμβρίου θα συζητηθεί το θέμα στην Ολομέλεια. Θα τα ξαναπούμε στις 2.30 ε, όπου έχουμε τη δημόσια ακρόαση με την Έλκε Κένικ, πρόεδρο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγείας. Σας ευχαριστώ.